So uh, um, Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας. Θα πάμε τώρα στα δύο θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα τα εξετάσουμε από κοινού. Θα μιλήσουμε για το κόστος της διαφθοράς στις αναπτυσσόμενες χώρες, πώς αποτελεσματικά χρησιμοποιείται η βοήθεια και για το επόμενο θέμα από κοινού. Οι δύο κύριοι θα μας παρουσιάσουν τα συμπεράσματά τους και μετά θα προχωρήσουμε στην άποψη της ΕΝΤΕΒΕ ε, σχετικά ε, με την καταπολέμηση της διαφθοράς ε, και συνέχιση το ψήφισμα της Ειδικής Επιτροπής ΚΡΙΜ. Κατά την παρουσίαση θα ενημερωθείτε και θα ακολουθήσει η συζήτηση. Η διαφθορά υποσκάπτει την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Έχουμε παράνομες ροές μέχρι ένα τρεις, εκεί εκτιμώνται οι παράνομες ροές και αυτά τα χρήματα αφορούν ε, τις αναπτυσσόμενες χώρες και τους φτωχούς ανθρώπους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταβάλει προσπάθειες να περιορίσει τη διαφθορά στις υποψήφιες χώρες ε, και στις ε, όμορες χώρες, αλλά δεν υπάρχει αρκετή πρόοδος ε, όσον αφορά τις σχετικές πρωτοβουλίες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έτσι λοιπόν έχει φτάσει στιγμή να ενισχυθούν τα συστήματα κατά τη διαφθοράς στις αναπτυσσόμενες χώρες. Με μεγάλη μου λοιπόν χαρά καλωσορίζω στην Επιτροπή μας τους δύο συντάκτες της έκθεσης. Ε, έχετε ε, τις ε, εισηγήσεις τους και των δύο εισηγητών ε, που είναι σύμβουλοι στο Ινστιτούτο Κρίσιαν Μίκελσεν της Νορβηγίας. Θα έλεγα λοιπόν να δώσουμε πρώτον λόγο στον Ιγνάτσιο Κοράο, ο οποίος είναι εισηγητής ε, για τη γνωμοδότηση. Μετά θα ακολουθήσει ε, μια εισήγηση για το ε, ξέπλυμα του, βόρου, του βρώμικου χρήματος που εγκρίθηκε από το ε, ψήφισμα και το οποίο περιλαμβάνει συστάσεις για δράση ε, στον αγώνα κατά της ε, διαφθοράς. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονές μας οι οποίοι θα παρουσιάσουν την έκθεσή τους 10 λεπτά ο καθένας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσουμε τα απορίσματα της μελέτης μας. Θέλω πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω με κάποια στοιχεία. Στοιχεία που περιλαμβάνει η μελέτη μας για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Όπως είπε και ο πρόεδρος, ε, η μελέτη διαπίστωσε ότι περίπου 1-3 δολάρια χάνονται κάθε χρόνο από παράνομες ροές ε, χρημάτων. Μία πρόσφατη μελέτη ε, μετά από μια σχετική πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε από το 2-3 μέχρι το 12 διαπιστώθηκε ότι χάθηκαν 6,63 που αφορούν στις αναπτυσσόμενες χώρες. 100 δις ε, δολάρια κάθε χρόνο ε, προσφέρονται σε τι σε βάση. Η βοήθεια αυτή για κάθε δολάριο που δίνεται 10 δολάρια φεύγουν με παράνομες ροές. Υπάρχουν κάποια στοιχεία για παράνομες ε, ε, ροές, ε, δεν υπάρχουν τόσο σαφή στοιχεία για τη διαφθορά. Φαίνεται όμως ότι το 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ χάνεται στην παγκόσμια διαφθορά και μεγάλο είναι το ποσό που χάνεται και από τους εθνικούς προπολογισμού λόγω της διαφθοράς. Καταλήγουμε λοιπόν στο ότι περίπου 20 μέσα τις, ε, το 40% των χρημάτων που δίδονται χάνονται. Στην μελέτη μα, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλέ δυσκολίε να μετρήσει κανείς το κόστος. Βεβαίω και μπορεί κανείς να αμφισβητήσει κάποιε από τις μεθόδου που χρησιμοποιούνται. Παρόλα αυτά, αν, τα στοιχεία, αν και τα στοιχεία δεν είναι ακριβή, διαπιστώνεται ότι αφορούν ε, μεγάλα ποσά και από την προοπτική των αναπτυσσόμενων χωρών βλέπουμε ότι αποτελούν πρόκληση για την ανάπτυξη αυτών των χωρών. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι επιπτώσεις είναι άμεσες, αλλά υπάρχουν στοιχεία ότι οι παράνομες ροές επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη. Επιπλέον, ε, μιλάμε για δυσαναλογία ε, αύξηση της ανισότητας. Ε, υποσκάπτονται οι δημόσιες υπηρεσίες. Υπάρχουν ε, απειλές για το περιβάλλον. Πολλά από αυτά τα θέματα πρέπει κανείς να τα έχει κατά νου. Βεβαίως μπορεί κανείς να πει ότι πολλά από αυτά θα προέκυταν και χωρίς τη διαφθορά. Όμως παράλληλα πρέπει να δούμε τι είδους ανάπτυξη θα μπορούσε κανείς να επιτύχει λόγω όλων αυτών των στοιχείων τι ε, θα μπορούσε επίσης να συμβεί αν την αφήσουμε ανεξέλεγκτη διαφθορά και αυτό πρέπει να το δούμε. Τα στοιχεία είναι καταθλιπτικά αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δικαιολογία για να απομακρυνθούμε από τις αναπτυσσόμενες χώρες και να πάψουμε να τους προσφέρουμε βοήθεια. Η απειλή παράνομων ροών και διαφθοράς ε, είναι μια απειλή για την ανάπτυξη και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα για να αντιμετωπιστεί η διαφθορά και για να φτάσει τελικά η βοήθεια στους δικαιούχους. Και θέλω να δώσω το λόγο στον Γέσπε, ο οποίος θα σας παρουσιάσει με ακρίβεια όλα αυτά τα θέματα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους και όλες για την πρόσκληση. Ε, ο συνάδελφος Νίλς σας είπε γιατί είναι σημαντική ε, γιατί είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τη διαφθορά και ότι η ευφιές είναι να καταπολεμηθεί η διαφθορά, γιατί, η διαφθορά γιατί αυτό σημαίνει πιο αποτελεσματική βοήθεια. Εγώ τώρα θα σας παρουσιάσω ως αναπτυξιακό ε, παράγον τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μετριάσει τη διαφθορά. Να αναλύσουμε επίσης ε, αν τα καταφέρνει καλά και να διεκπώσουμε συστάσεις για το τι παραπάνω μπορεί να κάνει. Το βασικό μήνυμα το οποίο θέλουμε σε αυτή τη σύνοδο να σας δώσουμε είναι ότι θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα και αυτό μάλιστα να αποφύγει προς όφελός της ε, και για τις ανεψόμενε χώρες βέβαια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μια συνεκτική στρατηγική για την πάταξη της διαφθοράς σε ανεψόμενε χώρες και να μελετήσει τα μέσα τα οποία θα είχε για την καταπολέμηση του φαινομένου εκτός των συνόρων τη. Τώρα, για τα επόμενα 10 λεπτά θα ήθελα να σχολιάσω τέσσερα σημεία. Το πρώτο είναι η ανάγκη ιεράρχησης προτεραιοτήτων, να δοθεί προτεραιότητα στο θέμα και η απαραίτητη πόρη. Το δεύτερο είναι ότι η στρατηγική προσέγγιση που ισχύει αυτή τη στιγμή δεν είναι επαρκής. Τρίτον, οι εταίροι που καλούνται να εφαρμόσουν έχουν επίσης σημαντικό ρόλο. Και τέταρτον, πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα κεραιότητας ε, στις χώρες εταίρους για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τον έλεγχο του φαινομένου. Το πρώτο θέμα λοιπόν για τις προτεραιότητες και τις επαρικές πόρους. Ίσως είναι και το πιο σημαντικό σημείο. Ω αναπτυξιακό παράγων, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει προτεραιότητα ε, στην αντιμετώπιση τη διαφθορά σε αναπτυσσόμενε χώρε και λίγη είναι η πόρη που διαθέτει για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Κατά την άποψή μα, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται εσωτερικά περισσότερη εμπειρογνωμοσύνη για να μπορεί να επιβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων, το πώς δαπανώνται τα χρήματα εκτός ε, ε της Ένωσης, να κάνει πιο πολλούς επιτόπιους ελέγχους, δέουσα επιμέλεια, ε, δειγματοληπτικούς ελέγχους, ε, σύστημα ε, πληροφόρησης, δηλαδή μετάλλευση πληροφοριών από πληροφοριοδότες, έναν κατάλογο ή καταλόγους για να βλέπουν ποια είναι τα προβλήματα. Όλα αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε λιγότερη διαφθορά ε, στα προγράμματα τα αναπτυξιακά. Υπάρχει μεγάλη αντίθεση μεταξύ της ε, σημασίας που δίνεται η καταπολέμηση στη διαφορά στις γειτονικέ χώρες έναντι των αναπτυσσομένων η φιλοδοξία και η αποφασιστικότητα που βλέπουμε σε ό,τι αφορά τι υποθέσεις υποθέσει και τη διαδικασία της διεύρυνσης δεν ε, φαίνεται να μεταδίδεται και να επεκτείνεται στην αναπτυξιακή βοήθεια παρά το ιστορικό. Ε, είχαμε δηλαδή πολύ φιλόδοξες ε, μεταρρυθμίσεις στις χώρες οι οποίες προσπαθούν φιλοδοξούν να γίνουν μέλη της Ένωσης, αλλά με τη στρατηγική που ακολουθείται σήμερα δεν εξετάζεται και το πώς θα μπορούσε να μειωθεί η διαφθορά στην αναπτυξιακή βοήθεια. Ε, συνάγουμε το συμπέρασμα ότι θα μπορούσε η Ένωση να ε, δώσει προτεραιότητα στον έλεγχο της διαφθοράς σε αναψώμενες χώρες και αυτό να βοηθήσει να δίνεται πιο αποτελεσματική αναπτυσσιακή βοήθεια. Δεύτερον, ανεπάρκεια της σημερινής στρατηγικής προσέγγισης. Θέλουμε να τονίσουμε ότι θα πρέπει ε, να δούμε το ιστορικό για να καταλάβουμε το υπόβαθρο, για να καταλάβουμε την κατάσταση. Η σημερινή σταδίκη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναπτύσσεται για τα κράτη-μέλη και για τις υποψήφιες προσένταξη χώρες. υποψήφιες χώρες και προσχωρούσες χώρες. Θα μπορούσε ε, να πει κανεί όμως ότι είναι πολύ λίγα αυτά που γίνονται για την αναπτυξική βοήθεια. Δεν αρκεί να βασίζεται κανείς στους ελέγχους. Ε, η στρατηγική δίνει έμφαση στους όρου, ε, στην αιρεσιμότητα. Δεν εξετάζει όμω ούτε εξηγεί σε βάθο πώ αυτό θα επηρέαζε και θα περιόριζε τι διαφθαρμένε συμπεριφορέ. Δεν εκπλήσει το ότι οι στρατηγικέ των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. πολύ λίγες αναφορές κάνουν ε, στη διαφθορά ή την καταπολέμηση της διαφθοράς για μερικές ουσιοδιαφθαρμένες χώρες στον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να στηρίξει τις προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς ενωση στις τρίτες χώρες, μη βασιζόμενοι μόνο όμως στους ελέγχους. Πρέπει να προωθηθούν μεταρρυθμίσεις ε, και ελπίζουμε ότι και η όρη, η αρεσιμότητα θα λειτουργήσει. Θα έπρεπε δηλαδή με άλλα εργαλεία καταπολέμησης πρόληψης διαφθόρας να συμπληρωθούν οι ε, και να ενισχυθούν οι μεταρρυθμίσεις και οι θεσμοί καταπολέμησης της διαφθοράς στις χώρες εταίρους. Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί σε στρατηγικές για έφραυστα, ε, ευάλωτα κράτη, παραδείγματος χάρη σε οποιοδήποτε μελλοντικό ε, πρόγραμμα για την ασφάλεια, για την ε, ανάπτυξη. Προτεραιότητα λοιπόν κοινή η ασφάλεια αλλά και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Το τρίτο σημείο, ο βασικός ρόλος των ε, εταίρων που αναλαμβάνουν την εφαρμογή που την υπεύθυνοι για την εφαρμογή. Θα πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικέ δικλείδε για την καταπολέμηση τη διαφθοράς που θα πρέπει να του υιοθετούν οι εταίροι του διάβλου. Γιατί ο αδύνατος κρίκος, ο αδύναμος κρίκος ε, δεν βρίσκεται στις ε, διαδικασίες της Ένωσης, ε, αλλά στην αντιμετώπιση καταστάσεων όπου τρίτα μέρη αναλαμβάνουν την εφαρμογή των πόρων, την, της βοήθειας. Βασίζεται σε τέρους όπως είναι και ο σάγια παράδειγμα η Ένωση για την υλοποίηση κάποιων προγραμμάτων εντός της Ένωσης ή σε χώρες που μπορούν, που επιθυμούν να προσχωρήσουν. Είναι αυτοί οι έμπιστοι εταίροι, όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν να προσφύγει σε αυτούς για την αναπτυξιακή βοήθεια. Υπάρχουν άλλοι πολυμερείς ε, δωρητές. Δεν μπορεί να ασκήσει δέος επιμέλεια παρακολούθηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ισχυρό εθνικό σύστημα ακαιρεότητα, όπως το λέμε, για την πάταξη της διαφθοράς. Η Ενώση πρέπει να εργαστεί πιο δραστήρια για να στηρίξει την ανάπτυξη ισχυρών εθνικών συστημάτων ακαιρεότητα, από τι χώρε που λαμβάνουν απτυξιακή βοήθεια. Γιατί βλέπουμε ότι δίνεται η βοήθεια αυτή ε, από την Ένωση μέσω των εταίρων εφαρμογή υλοποιείται, ε, μπορεί να δίνεται και δημοσιονομική στήριξη. Αλλά δεν υπάρχει επαρκή στελέχωση για το σύστημα κεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μαζί με άλλου, θα έπρεπε να βοηθήσει να δημιουργηθούν ισχυρά τοπικά συστήματα για τον έλεγχο τη διαφθορά, δηλαδή μιλάμε για την κεντρική κυβέρνηση και για τι ε, τοπικέ αρχέ, ανοιχτοί προπολογισμοί, διαγωνισμοί και μηχανισμοί λογοδοσία ώστε να μπορούν να επαγρυπνούν και φορεί και πολίτες ε, για τον έλεγχο τη διαφθοράς. Λίγα γίνονται όμω σε σχέση με το συνολικό όγκο της διατηθέμενη βοήθεια. Ε, συνόψη. Ω πρώτο συμπέρασμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ω αναπτυξιακό φορέα ε, βρίσκεται, υπολείπεται άλλων αντίστοιχων παράγοντων η Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά την αντιμετώπιση τη διαφθορά. Χρειάζονται περισσότεροι επιτόπιοι έλεγχοι, δειγματοληπτικοί έλεγχοι, ένας κατάλογος είπαμε, checklist και προσπάθεια ώστε οι πρωταθλητές ακεραιότητας που θέλουν την υποστήριξη να την έχουν αυτή την υποστήριξη. Και αυτό θα οδηγήσει κατά πάσα πιθανότητα σε λιγότερη διαφθορά. Οι συστάσεις μας λοιπόν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι Ελπίζουμε να ξεκινήσετε μια διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικής ε, που θα ε, ξεκαθαρίσει ποια είναι η θέση της Ένωσης για τη διαχείριση του κινδύνου της διαφοράς ιδίως στις αναψώμενες χώρες, να αναγνωριστεί ότι πρέπει ε, να βελτιωθούν τα συστήματα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, να ενισχυθούν δυνατότητες, ικανότητες των εταίρων για των εφαρμοστικών φορέων και των εθνικών εποπτικών αρχών. Επίσης, ελπίζουμε να εξετάσετε το κόστος, τη σχέση κόστος ωφέλους ε, της σημερινής στρατηγικής και το κατά πόσο υπάρχει στελέχωση ε, των φορέων για την αντιμετώπιση της διαφθόρας. Να δημιουργηθεί μια άλλη προσέγγιση ε, ολοκληρωμένη που είναι κατακαιρματισμένη αυτή τη στιγμή σε επίπεδο κυβερνητικό για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Επίσης, καλό θα ήταν να καταρτιστούν κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση περιστάσεων κινδύνου, οι εταίροι που ε, είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή να έχουν ε, τους μηχανισμούς του καταπολέμησης της διαφθοράς ε, και τη δυνατότητα να περιορίσουν το φαινόμενο αυτό όσο το δυνατό περισσότερο. Η δημοσιονομική στήριξη θα πρέπει να συνοδεύεται επίση από, βασικά, από συγκεκριμένα σχέδια για το μετριασμό των κινδύνων και θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται οι προσπάθειες πάταξης της διαφθοράς και χρήσιμο θα ήταν να δοθεί καλύτερη επιχειρησιακή καθοδήγηση με τη χρήση της αιρεσιμότητας ε, για αντιμετώπιση περιπτώσεων διαφθοράς και για να αναλυθούν πολιτικές δεσμεύσεις. Τέλος, θέλουμε να τονίσουμε ότι ελπίζουμε να συνεχίσετε την ε, καλή πρόοδο εξασφαλίζοντας ε, την χρηματοοικονομική ροή με νέες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση ε, των ε, δημόσιων διοικήσεων μπορούν να ελέγχουν τα φαινόμενα φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής, διαφθοράς και επίσης καλύτερη διεθνή συνεργασία για να μην ε, υπάρχουν πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Ευχαριστώ. Okay. Thank you both for the... Σας ευχαριστούμε και τους δύο για τις παρουσιάσεις αυτές και για την έκθεσή σας. Μπορεί τώρα να ξεκινήσει η συζήτησή μας και θα δώσω καταρχάς το λόγο στον Ιγνάτσιο Κοράο ο οποίος είναι εισηγητής μας. Σας παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ καταρχάς να ευχαριστήσω τους δύο προσκεκλισμένους μας που πήραν το λόγο για αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία μας δώσατε. Έχουμε εδώ πέρα μια πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων βάσει βέβαια ενός κειμένου που δεν έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας δεν έχουμε ακόμα την έκθεση στα χέρια μας, επομένω κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για ένα ζήτημα το οποίο το είπατε κι εσείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς στα πλαίσια άλλων εκθέσεων, όπως για παράδειγμα στην έκθεση που είχαμε κάνει για την φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή ή στα πλαίσια μιας άλλης έκθεσης για την χρηματοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης των απτυσσομένων χωρών, είχαμε αναφερθεί στο ζήτημα της διαφθοράς. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε 1-3 ευρώ ετησίως και για το ότι πολλές φορές για κάθε 1 ευρώ το οποίο δίνουμε σε μια αναπτυσσόμενη χώρα μας διαφεύγουν 10 ευρώ στα χέρια της διαφθοράς των διαφθαρμένων δικτύων. Νομίζω λοιπόν ότι το ζήτημα της διαφθοράς πραγματικά θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο των συζητήσεών μας κάθε φορά που μιλάμε για αναπτυξιακή βοήθεια και αναπτυξιακή χρηματοδότηση. Είναι σαφές ότι η διαφθορά πραγματικά αποτελεί τροχοπέδι στην οικονομική ανάπτυξη των απτυσσόμενων χωρών και πλήττει ιδιαίτερα τους πιο φτωχούς ανθρώπους. Στην έκθεση λοιπόν αυτή την οποία θα συντάξουμε προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, στην γνωμοδότησή μας δηλαδή, θέλουμε να ασχοληθούμε με διάφορα ζητήματα και μας δίνεται αυτή τη στιγμή μια καταπληκτική ευκαιρία για να ξεκινήσει μια κάποια συζήτηση. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια, ένας πολύ στενός σύνδεσμος ανάμεσα στη διαφθορά την παγκόσμια κυβέρνηση, καθώς επίσης και διάφορα δίκτυα τα οποία βάλουν κατά του περιβάλλοντος. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε καταρχάς ποια είναι η σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε κάποιες πλούσιες χώρες, οι οποίες εκμεταλλεύονται πιο φτωχέ χώρε και πειράζουν βέβαια και την οικονομική βοήθεια που δίδεται στις χώρες αυτές. Ας μην ξεχνάμε επίση ότι η διαφθορά μπορεί να καταλήξει να χρηματοδοτεί ακόμα και την τρομοκρατία και νομίζω ότι αν είχαμε καλύτερα περιβαλλοντικά κριτήρια θα μπορούσαμε να προτείνουμε κάποια πιο αυστηρά πρότυπα όσον αφορά την παροχή της ε, αναπτυξιακής βοήθειας. Νομίζω ότι θα πρέπει το ζήτημα αυτό να μπει στο κέντρο πραγματικά της ε, ατζέντας που έχουμε για την αναπτυξιακή βοήθεια για το έτος 2015 και για τα επόμενα έτη. Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα καλύτερα παραδείγματα που έχουμε σε εθνικό και διεθνέ επίπεδο όσον αφορά την καταπολέμηση τη διαφθορά. Έχουμε και κάποια παραδείγματα θετικά, όχι μόνο στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε και κάποια εθνικά μέτρα τα οποία έχουν εγκρίνει χώρε όπω η Λιβερία Κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε και τη δική μας τη θέση και βέβαια έχουμε και κάποιες διεθνείς συμβάσεις που έχουν συμβάλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στην καταπολέμηση των παράνομων οικονομικών ροών. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να εγκρίνουμε όλο και περισσότερα τέτοια μέτρα με διεθνή εμβέλεια. Θα πρέπει όμως να καταφέρουμε να ενισχύσουμε και την κοινωνία των πολιτών καθώς επίσης και την χρηστή διακυβέρνηση για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και κατά αυτόν τον τρόπο περνάω στο τέταρτο σημείο που έθεσε ο κύριος Τζόνσον, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα διακυβέρνηση και τα μεμονωμένα κράτη-μέλη με τα οποία εμείς έχουμε σχέση ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Να καταφέρουμε δηλαδή να βοηθήσουμε την διοίκηση των χωρών αυτών να καταπολεμήσει τη αυθορά, αρκεί βέβαια να υπάρχει μια αρχική θετική βούληση αυτών των κρατών. Νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να ασχοληθούμε και με το ζήτημα της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή πάλι να βρούμε αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να δημεύσουμε, να κατασχέσουμε περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτελούν έσοδα προϊόντα τελικά εγκληματικής δραστηριότητας. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το κάνουμε καλά-καλά ούτε στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπο αποτελεσματικό. Έχουμε κάποιες νομοθεσίες σε κάποια κράτη-μέλη κατά της διαφθοράς που είναι πιο ανεπτυγμένε σε σχέση με άλλες νομοθεσίες. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να δώσουμε εμεί μαθήματα ω Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να συμβάλλουμε με τρόπο φιλόδοξο προκειμένου να καταφέρουν και τρίτε χώρε, αναπτυσσόμενε χώρε, να καταπολεμήσουν τη διαφθορά. Αυτό είναι στόχο άλλωστε και τη έκθεση που θα συντάξει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Χρειάζεται καλύτερη αμοιβή εμπιστοσύνη, συνεργασία δικαστικών αστυνομικών υπηρεσιών, καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών, βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, καλύτερο πλαίσιο όσον αφορά τι ποινικέ έρευνε. και οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα συστήματα προστασίας των μαρτύρων, των πληροφοριοδότων, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό κριτήριο για να καταφέρουμε να συνεργαστούμε με ορισμένες χώρες για την καταπολέμηση πολλών μορφών εγκληματικότητας. Καλύτερη χρήση τώρα των διαφόρων ταμείων και πόρων που έχουμε. Ξέρετε ότι μιλάμε πολλές φορές για το 20 ή 40% πολλές φορές όσον αφορά, όταν μάλλον ένα 20 με 40% της αναπτυξιακής βοήθειας μπορεί τελικά να περάσει στα χέρια της μαφίας ή εγκληματικών οργανώσεων, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε όντως να αγγιόμεθα, να διασφαλίζουμε ότι όντως τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούνται για την απτυξιακή βοήθεια, ότι όντως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία θα ωφελήσουν επιτόπου τις χώρες και τους πληθυσμούς τους. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε μια επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, ιδίω εν ώψη του εγγράφου αυτού που πρόκειται να συντάξω. Η διαφθορά έχει να κάνει βέβαια και με τη διαφάνεια, καλύτερη διαφάνεια στην διακυβέρνηση, καλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και να καταφέρουμε τελικά να εγκαθιδρύσουμε περισσότερο σε κάποιες χώρες το κράτος δικαίου. Νομίζω ότι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και γενικά πρέπει να επικεντρωθούμε τρία αυτά στοιχεία τα οποία έθιξε. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε. Τώρα λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ε, ε, ε δεν είναι εδώ ο σκιώδης του ΕΛΚΑ, αλλά των σοσιαλδημοκρατών. Βεβαίως, αν επιθυμεί και κάποιος άλλος από το ΕΛΚ να λάβει το λόγο, ε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και όλους όσοι παρουσίασαν αυτά τα πολύ σημαντικά στοιχεία και χρήσιμα για τη δουλειά του συναντέλφου Κοράου και τη δική μας δουλειά που είμαστε ισκιώδεις εισηγητές. Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή σχέση ανάμεσα στη μάχη κατά της διαφθοράς και την ενίσχυση ε, της ε, λογοδοσίας εναντί των πολιτών να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Ε, είναι σημαντικό να υπάρχει χρηστή διαχείριση στο καινούριο πλαίσιο μετά το 2015 επιτέλους ε, θα υπάρχει και ένα νέος στόχος που θα αφορά την good governance την ε, καλή διακυβέρνηση αλλά και ε, την λογοδοσία, τη διαφάνεια και τον αγώνα κατά της διαφθοράς. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Και εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, το εξής. Κατά πόσο γνωρίζουμε τη σημασία των ε, δικτών. Ε, να μπορεί κανείς να μετρήσει. Γιατί για κάθε ένα από τους στόχους που ορίζονται θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορούμε τελικά να μετρήσουμε την καλή διακυβέρνηση που είναι δύσκολο να μετρηθεί κυρίως όσον αφορά τον αγώνα κατά της διαφθοράς. Η διαφθορά έχει άμεση επιπτώσει στην ανάπτυξη, στη βοήθεια, στη δυνατότητα να ε, προμηθεύονται οι δημόσιες υπηρεσίες. Αν θέλετε και όσον αφορά την ανισότητα, πρέπει να οριστεί η διαφθορά ε, σαν ένα είδος ε, φόρου τον οποίο πληρώνει το πιο ευάλωτο κομμάτι της κοινωνίας, αναδρομικού φόρου. Και νομίζω ότι θίξατε και ένα πολύ σημαντικό θέμα, επί του οποίου την προηγούμενη εβδομάδα μόλις ψηφίσαμε ε, το θέμα των παράνομων οικονομικών ε, ροών και της ε, φόρου διαφυγής που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διαφθορά. Τιμήσατε τις διαστάσεις του φαινομένου που είναι τεράστιες και με τον τρόπο αυτό υπάρχει κίνδυνος ε, να είναι ανεπαρκής οι δικές μας οι δομές αν δεν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί αν δεν τα καταφέρουμε με το ένα χέρι θα ε, παίρνουμε ό,τι προσπαθεί να δώσει το άλλο. Το ψήφισμα το οποίο ψηφίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, εκεί ζητάμε την πλήρη Φάνια όσον αφορά τους ε, τελικούς αποδέκτες. Και αυτό για να αποφύγουμε να υπάρχουν ε, εταιρείε ε, φάντασμα, ένα δίκτυο τέτοιων εταιρείων που θα αποκρύπτουν χρήματα που προέρχονται από τη διαφθορά και από την παράνομη οικονομία από παράνομες οικονομικές ροές, ακόμα και από τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτό ανέφερε ο συνάδελφος. Άρα δηλαδή θεωρώ ότι η διαφάνεια είναι το πιο αποτελεσματικό αντίδοτο που έχουμε στη θέση μας και πρέπει να το προβάλλουμε περισσότερο. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν ε, εργαλεία σε διεθνές επίπεδα και υπάρχουν αυτά, όπως μια διεθνωτή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια. Θα ήθελα όμως να γνωρίζω ποια είναι η εμβέλεια αυτών των διεθνών οργανώσεων. Ε, στο στόχο υπαρτημών 16 γίνεται λόγος και γι' αυτό. Οι χώρες, οι αναπτυσσόμενες χώρες πώς συμμετέχουν στη συζήτηση και πόσο. Παραδείγματο χάρη οι χώρες αυτές συμμετέχουν περισσότερο και στα ε, αντιφατικά εργαλεία συμμετέχουν σε ένα πραγματικό οργανισμό, διότι δεν μπορούμε να έχουμε κατά νου να αναπτύξουμε αποτελεσματικά εργαλεία χωρίς ε, να υπάρχει άμεση συμμετοχή ε, και των ε, οργανισμών και των εμπειρογνωμόνων. Τελειώντας θα ήθελα να πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όταν θα είναι έτοιμη η εισήγηση. Θα έχουμε ακόμα πολλά να πούμε και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι το εξή. Πολλές φορές υπάρχει διαφθορά και στην προσπάθεια να προσελκύσει κανείς ε, ε, επενδύσεις από αναπτυγμένες χώρες. Ε, συμφωνίες που βασίζονται σε κίνητρα για φοροαποφυγή. Και αυτά αποδεικνύονται ιδιαίτερα επικερδή για τις εταιρείες αλλά όχι για τις χώρες. Και γι' αυτόν λοιπόν το λόγο και κάτω από αυτό το πρίσμα εμείς επιθυμούμε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και να εφαρμόζονται ε, κάποια συγκεκριμένα εργαλεία όπως ανταλλαγή απόψεων, ε, εκθέσεις αναχώρα και παρεμφερή. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος κοιόδης, ε, οπότε το λόγο μπορεί να πάρει οποιοδήποτε άλλος συνάδελφος θέλει το λόγο από πολιτικές Τσέλερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για τη μελέτη που εκπονήσατε και για την ε, εισήγησή σας. Διαβάζοντας βέβαια τη μελέτη, πραγματικά ε, απογοητεύεται κανείς. Γιατί τα παραδείγματα τα οποία αναφέρετε είναι εκείνα όπου έχουμε κάποιες ε, ε, υποψίες, αλλά εσείς ε, τα παρουσιάζετε ξεκάθαρα. Και αυτό κυρίως εκεί που γίνεται λόγος για την βοήθεια που χορηγείται, λέτε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, σαφείς οδηγίες ε, για την καταπολέμηση της διαφθοράς, κάτι το οποίο πολλές φορές είναι θύμα άλλων προτεραιοτήτων. Πολλές φορές είμαστε αναγκασμένοι να ε, συνεργαζόμαστε με κάποιες χώρες για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας ή αν θέλετε για την αντιμετώπιση κρίσεων και παρεμφερών και εκεί ακριβώς σε αυτόν τον αγώνα εμφανίζονται πράγματα που ε, θα έπρεπε να τα προβάλλουμε καλύτερη δηλαδή διακυβέρνηση, ε, καλύτερη, μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτά όμως μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Ε, και εξαιρετισμενοι αυτό. Γυρίζουμε γύρω γύρω από την ουρά μας. Και πού είναι η λύση το σύστημα των χρηματοδοτικών ροών είναι αποτελεσματικό. Μήπως πρέπει να αναζητήσουμε άλλες λύσεις όπου θα είμαστε καλύτερα προστατευμένοι, θα είμαστε πιο σίγουροι. Θα είμαστε πιο σίγουροι ότι τα χρήματα τα οποία στη τελική ανάλυση ε, χρειαζόμαστε για τη βελτίωση της κατάστασης στις ενδιαφερόμενες χώρες, τα χρήματα αυτά να φτάνουν πραγματικά στον τελικό αποδέκτη και όχι στις τσέπες κάποιων λίγων που ε, απλά πλουτίζουν παραπάνω. Η κυρία Χόιμπουχ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε πολύ και για τη μελέτη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι για άλλη μια φορά φαίνεται πόσο σημαντικό είναι να προσπαθεί κανείς να δει το κατά πόσον τα χρήματα που διαθέτουμε φτάνουν στον επιθυμητό τελικό αποδέκτη. Εσείς το αναφέρετε ότι ε, τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει ε, παρακολούθηση, αξιολόγηση. Τι γίνεται τελικά με τα χρήματα αυτά. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ήδη είπατε εσείς. Ε, σε πάρα πολλά σημεία είπατε ακριβώς ε, που ήθελα να πω και εγώ. Εγώ ήθελα να μιλήσω για την φοραποφυγή, για παράνομες οικονομικές ροές το είπε και ο συνάδελφος ότι χωρίς ε, την διαφθορά δεν έχουμε τις ε, παράνομες ροές και οι παράνομες ε, ροές είναι εκείνες που επιτείνουν τη διαφθορά αλλά φοβάμαι ότι και στην Ευρώπη δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Δηλαδή μιλάμε για φοροαποφυγή και πολύ συχνά πρόκειται για θέματα τα οποία λαμβάνουν χώρα σε πολυεθνικό επίπεδο. Και έχουμε πολλές ε, πολυεθνικές επιχειρήσεις και χρήματα τα οποία επενδύονται σε πολυεθνικές και δημιουργείται λοιπόν πρόσφορο έδαφος για φοροαποφυγή. Ε, αυτό ε, ας μην ξεχνάμε ότι είναι έγκλημα γιατί αφορά τα χρήματα του δημοσίου. Δεν είναι ένα απλό πλημέλημα. Γίνεται λόγος για διαφάνεια. Σημαντικό αυτό, αλλά κάτι που επίσης είναι σημαντικό, είναι πολιτική βούληση. Είπατε ότι μετατοπίστηκαν οι προτεραιότητες. Αυτό μερικές φορές μπορεί να συμβαίνει λόγω κάποιων αναγκαιοτήτων. Αλλά αυτό που παίζει ρόλο είναι να βλέπει κανείς ε, το γενικότερο πλαίσιο. Και όταν μετατοπίζονται οι προτεραιότητες ε, σε κάποιους τομείς. Όταν όμως έχουμε κατά νου την διαφθορά πρέπει να γνωρίζουμε ότι μετατοπίζονται και οι οικονομικές ροές φτάνουν σε λάθος χέρια. Άρα ε, πολιτική συνέπεια πρέπει να επιδεικνύεται γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος και η άλλη είναι ότι στην Ευρώπη θα πρέπει να τα δούμε λιγάκι κάπως καλύτερα τα πράγματα, ε, να δεσμεύσουμε τις δικές μας τις χώρες, να μιλήσουμε ε, για τους προλογικούς παραδείσους και αν εμείς δεν τα κάνουμε καλά, πώς μπορούμε να καλούμε τις άλλες χώρες να έχουν ακέραια χρηματοδοτικά και φορολογικά συστήματα. Και είναι απαραίτητο να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών ε, να υπάρχει αυτή η έκθεση αναχώρα. Εάν το φορολογικό απόρριτο το διατηρούμε, πώς ε, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά. Όλα αυτά πρέπει να τα επιτύχουμε σε διεθνές επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι οι επιχειρήσεις μας ε, έτσι και αλλιώς δουλεύουν σε διεθνές επίπεδο και έτσι αν δεν ε, συνεργαστούμε νομίζω ότι θα είμαστε αναγκασμένοι να τρέχουμε συνέχεια πίσω από τις επιχειρήσεις και δεν θα ε, σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Χρειαζόμαστε και δεσμευτικούς κανόνες για την ε, ονομαζόμενη εταιρική ευθύνη και μόνο τότε μπορούμε, θα μπορούμε να μιλήσουμε για διαφάνεια όταν δηλαδή θα υπάρχει η πολιτική βούληση να αντιμετωπιστούν τα πράγματα επί της ουσίας. Σας ευχαριστούμε. Λόλα Σάντζες παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η διαφθορά έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη, ιδίω στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα πρέπει να δούμε πού οφείλονται αυτές οι δραστηριότητες και τι αποτελέσματα έχουν. Σίγουρα η διαφθορά, ιδίω ε, την Εφημερία των πολιτών πλήττει, δημιουργεί προβλήματα κυβερνητική αστάθεια, γιατί κανένα πολιτικό κόμμα δεν περιλαμβάνει ε, στο εκλογικό του πρόγραμμα την καταπολέμηση τελικά της διαφθοράς, άρα υπάρχει συνεχής απογοήτευση και αποστασιοποίηση τη κοινής γνώμης από τους πολιτικούς. Τους θεωρούν τελικά ε, πηγές προβλήματος και όχι επίλυσης προβλημάτων για τους πολίτες. Και αυτό είναι τελικά πρόβλημα για τη δημοκρατία και τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού σε πολλές χώρες. Η θεσμική διαφθορά επίσης <clears throat> έχει ως αποτέλεσμα να προωθούνται προγράμματα που ευνοούν την, ε, το χρηματισμό των πολιτικών και όχι την ε, βελτίωση του ιδιωτικού επίπεδου και πλήττεται πάντα ο πιο προστάτευτος πληθυσμός. Δημιουργείται επίση μεγαλύτερη γραφειοκρατία, διότι επιλέγονται υπάλληλοι για τη σιωπή του, ε, για την συνενοχή του και όχι για τι ικανότητέ του. Και αυτό πλήττει για μια ακόμα την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και κάτι άλλο, για το οποίο δεν γίνεται συχνά λόγο. Διαφθορά σε σχέση με τον περιορισμό θεμελιωδών ελευθερών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παραδείγματο χάρη, ελευθεροτυπία, δικαίωμα του ε, συνέρχεστε, του διαδηλώνει, και τώρα σε ό,τι αφορά τα αίτια της διαφθοράς, ιδίω σε αναπτυσσόμενες χώρες, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η κρατική ε, οικονομική δομή. Αν δεν υπάρχει διανομή του πλούτου, τελικά ε, έχουμε τη δημιουργία μιας οικονομικής ελίτ η οποία παγιώνεται και επίσης επηρεάζει και ε, κυριαρχεί και στο πολιτικό, στο πολιτικό στίβο. Πρέπει λοιπόν ε, να καλυφθούν πρώτα οι βασικές πρωταρχικές ανάγκες ε, του πληθυσμού γιατί αν δεν είναι αυτές οι ανάγκες καλυμμένες δύσκολα θα ασχοληθεί με την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς. πρέπει να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη, πρέπει να υπάρξει ισομερής κατανομή του πλούτου με τη σωστή φορολογική πολιτική. Γιατί μπορεί να κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δεν πιστεύουμε στην αιρεσιμότητα, στην αναπτυξιακή βοήθεια με βάση τα κριτήρια αυτά, γιατί αυτό θα δημιουργήσει μόνο προβλήματα στον πληθυσμό. Ούτε πάβει ε, η διαφθορά τελικά. Και αν συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο η κατάσταση, η χώρα μου, η Ισπανία και άλλες χώρες δεν θα παίρνουν ε, κονδύλια, διότι έχουν, δεν θα έπρεπε να παίρνουν κονδύλια, γιατί ε, πολλά κόμματα στη, και τα κόμματα της εξουσίας στην Ισπανία είναι διεφθαρμένα και λόγω της διαφθοράς ε, απειλείται η ευημερία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε συνεπείς στην εξωτερική πολιτική και ιδίω στην εμπορική πολιτική γιατί πολλές φορές υπάρχει συνενοχή μεταξύ ε, της ε, εμπορικής πολιτικής και των διαφερμένων ελίτ τρίτων χωρών. Και το βλέπουμε κατά την υπογραφή εμπορικών συμφωνιών. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ε, τότε η διαφθορά, μας ενδιαφέρει να βγάλουμε λεφτά και να βάλουμε χέρι στους φυσικούς πόρους για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ε, πρέπει όμως να δούμε τελικά ποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση εποφελείται από την ύπαρξη διαφθορά στις τρίτες χώρες και βέβαια αυτό το οποίο έλεγε η Έλλη πριν οι εταιρείε μας που είναι και σπεσιαλίστε στην, καταπολέ... στην φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή, ιδίω στι τρίτε χώρε. Επομένω, ε, ωραία είναι να το θέτουμε αυτό το ζήτημα και να μιλάμε για, για τα θέματα αυτά υπό το αναπτυξιακό πρίσμα και στην ε, Επιτροπή ΙΝΤΑ, ε, διεθνού, Υπουργού, να μην γίνεται λόγο για όλα αυτά τα θέματα τη διαφθορά. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον τέλο να αναπτυχθεί μια πρόταση ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει για την πρόθεση της αυτονομίας και ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος των αναπτυσσόμενων χωρών, κάτι που είναι κλειδί για την καταπολέμηση της διαφθοράς, πάντα βέβαια με την τήρηση συγκεκριμένων κριτηρίων. Ευχαριστώ. Okay, thank you, Mr. Neuser. <clears throat> Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές μας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θέλω όμως να προτάξω το εξής. Δεν πρέπει να συζητάμε με βάση το ότι από την μια πλευρά έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ασχοληθούμε ε, με το να περιοριστεί η διαφθορά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε τη δική μας θέση. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι κάθε χρόνο ένα εκατομμύριο ευρώ χάνεται λόγω της ε, φοροδιαφυγής μέσω φορολογικών παραδείσων και ε, λαθρέα εργασία. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρόβλημα. Και αν θέλουμε οι άνθρωποι στην Ευρώπη να έχουν κάποια προοπτική, οι άνθρωποι επιθυμούν το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί ενεργά, να προσφερθούν λύσεις, Για τελειώς θεωρώ ότι σε Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχουμε προοπτική. Τώρα, στο διατάφτα. Τα χρήματα των ε, φορολογουμένων πρέπει να ελέγχονται εκεί που φτάνουν. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και γνωρίζουμε ότι παντού υπάρχουν ε, κανονισμοί. Το ερώτημα είναι τι κανόνες υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ε, εντολές που έχουν δοθεί στην Κομισιόν, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όμως Θέλω να σα ρωτήσω λιγάκι γιατί δεν έχω καταλάβει αυτέ τι εντολές ή τι οδηγίε. Παραδείγματο χάρη λέτε ότι πρέπει να ενισχυθεί ο έλεγχο τη διαφθοράς. Χρειαζόμαστε πυρογάμους. Εντάξει, αυτό είναι συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο είναι επίση και το σύστημα των ε, καταγγελόντων, των whistleblowers. Ε, πρέπει όμω ε, να υπάρχει διαχείριση κινδύνου. Αυτό δεν το καταλαβαίνω καλά, να μας το εξηγήσετε λιγάκι. Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η διαφθορά γιατί με τον τρόπο αυτό ή από εκεί εξαρτάται και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όσο υπάρχουν διεφθαρμένοι άνθρωποι δεν υπάρχει ε, σταθερότητα και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η ακραία φτώχεια. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα στα κράτη και τα κράτη που θίγονται μόνα τους να αγωνίζονται για μεγαλύτερη αξιοπιστία. Υπάρχουν τέσσερις τομείς ε, που ήθελα να δείξω όσον αφορά την ε, υποστήριξη του προϋπολι... μέσω προϋπολογισμού ε, πολλοί μας λένε ότι μέσα από εκεί η διαφθορά είναι πολύ πιο εύκολη δηλαδή ε, τα ευρωπαϊκά μας γραφεία στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν το απαραίτητο όπλο για να αποκαλύψουν περιπτώσεις διαφθοράς. Και λέγεται και ότι όταν πρόκειται για κονδύλια που έρχονται από τον ε, προπολογισμό ε, είναι λιγάκι ανεκτική. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε λιγάκι το θέμα αυτό στις αναπτυσσόμενες χώρες και το θέμα του τύπου υπάρχει κάποιο απλοστάσιο για να αποκαλύπτονται αυτές οι περιπτώσεις. Και στην Ευρώπη υπάρχει διαφθορά, όμως ο τύπος βοηθάει να αποκαλύπτονται οι σχετικές περιπτώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις ΜΚΟ. Δηλαδή κατά πόσον οι ΜΚΟ μπορούν να αναλάβουν αυτό το ρόλο στις αναπτυσσόμενες χώρες και επίσης αυτό που παίζει ρόλο είναι κατά πόσον στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, που να είναι ε, κατά πόσο στις αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχουν τα απαραίτητα δίκτυα για να περιορίσουν τη διαφθορά. Σας ευχαριστούμε. Δύο ακόμα έχουμε, Γκέρενς και Χάουταλα. Ο Τσάρλς Γκέρενς πρώτος παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις έχω και μία παρατήρηση. Πρώτη ερώτηση. Όσον αφορά την αρεσιμότητα και τις προϋποθέσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί ένα σύστημα αιρεσιμότητας το οποίο είναι καλά ανεπτυγμένο δεν δίνει χρήματα αν δεν έχει διασφαλίσει ότι ακολουθούνται συγκεκριμένε πρακτικές από τους δικαιούχους. Άλλοι εταίροι όμως πάλι δεν είναι τόσο αυστηροί όσο εμείς και δεν έχουν καμία προϋπόθεση, κανένα σύστημα αιρεσιμότητος. Συνεπώς, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε ποτέ τη διαφθορά σε μια χώρα εταίρο, όταν η χώρα αυτή είναι εταίρος και με άλλες τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, οι οποίοι ενδεχομένω να ενθαρρύνουν τη διαφθορά, είναι οι ίδιες διαφθαρμένες. Πώς μπορούμε στην περίπτωση αυτή να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση, τι κάνουμε τις χώρες αυτές, τι προβλέπετε για τις χώρες αυτές και πώς θα πρέπει, ποια θα πρέπει να είναι η στάση που θα η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε αυτές τις χώρες. Για παράδειγμα, δίνουμε πιστώσεις, δίνουμε ένα δάνειο σε μια χώρα το οποίο η χώρα αυτή δεν το αποπληρώνει, αλλά παρόλα αυτά ε, καταφέρνει να εξασφαλίσει κάποια δικαιώματα εξαγωγών. Νομίζω ότι μιλάμε ουσιαστικά για ένα σύστημα διαφθοράς. Εμείς δεν θα το επιτρέπουμε ποτέ αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μία παρατήρηση. Ας μην είμαστε υποκριτές. Βλέπουμε γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν φτάσουμε σε ένα επίπεδο πλέον ανάπτυξης μπορούμε να επιβάλλουμε κάποια πράγματα απευθείας στους ε, εταίρους μας. Ενώ και εμείς οι ίδιοι χρειάζεται να καταβάλουμε πολλές φορές πάρα πολλές προσπάθειες μακροχρόνιες προκειμένου να φτάσουμε στην επίπεδο ανάπτυξης. Δεν μπορούμε αυτό το επίπεδο ανάπτυξης να το μεταφέρουμε αυτούσιο, αυτόματα σε μια χώρα εταίρο. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε μία στοχοθετημένη στρατηγική προσέγγιση προς τις χώρες εταίρους. Τέλος, φορολογία και διαφθορά. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν μια φορολογική νομοθεσία που καθιστά κάθε φορολογούμενο υπόχρεο απέναντι στις ε, Αμερικανικές φορολογικές αρχές. Ακόμα και αν δεν ε, κατοικεί ο φορολογούμενος αυτός στις Ηνωμένες Πολιτείες, οφείλει να κάνει δήλωση φορολογική στην Αμερικανική εφορία. Δεν θα μπορούσαμε κι εμείς κάτι αντίστοιχο να προτείνουμε σε όλες τις δικές μας τις χώρες Κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα προστατευόμασταν ε, από τη διαφθορά, από τα φαινόμενα διαφθοράς θα προστατεύαμε και εμείς τους ίδιους τους πολίτες μας αλλά και τους πολίτες των χωρών εταίρων μας. Κατά αυτόν τον τρόπο θα διευρύναμε ουσιαστικά το πεδίο δραστηριοποίησης των δικών μας φορολογικών αρχών και δεν θα επιτρέπαμε κατά αυτόν τον τρόπο στο να εμφανιστούν φαινόμενα διαφθοράς. Θα είχαμε δηλαδή, αν θέλετε, ένα δίκτυο ασφαλεία και προστασία από τη διαφθορά, το οποίο θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό. Uh, Ευχαριστώ και τελευταία η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. πολύ ευγνώμων για τη μελέτη που ακούσαμε πριν αρχίσει η συζήτηση και ευτυχώς που δεν είναι πια ταμπού στις, στον αναπτυξιακό διάλογο το θέμα της διαφθοράς, γιατί μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν. Είναι σαφές βέβαια ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε διαφθορά, δεν θα πρέπει να αυταπατώμεθα, γι' αυτό και η Κομισιόν ήδη από πέρυσι ε, εκπώνησε έκθεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι ένας σταθμός. Όμως το βασικό είναι ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον δεν αξιοποιούμε τα μέσα ε, που έχουμε στη διάθεσή μα ή δεν τα χρησιμοποιούμε επαρκώ για να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Αναφέρθηκε τη δημοσιονομική στήριξη. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη τον σημερινό ορισμό της δημοσιονομικής στήριξης. Δηλαδή συμβάσεις ε, ή συμβόλαια χρηστής διακυβέρνησης. Αυτό είπε ακριβώς ε, ο Επιτρόπος Πίμπαλξ όταν εθετήθηκε το 2012 αυτή η νέα έννοια. Τώρα κατά πόσον μιλάμε για γενική ή για τομεακή δημοσιονομική στήριξη, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μιλάμε για συμβάσει χρηστής διακυβέρνησης. Θα ελπίζω ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις άλλες ε, καλές πρακτικές ε, για να χρησιμοποιήσουμε ε, αυτά τα μέσα για, ως μοχλό, ως μόχλευση για χρηστή διακυβέρνηση θα μπορούσαμε να έχουμε ίσως συνεργασία με άλλους ε, χρηματοδότες. Και εκεί που είναι σημαντικό χρηματοδότηση η Ένωση και είναι συχνά, θα πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της διαφθοράς, με τη βοήθεια της δημοσιονομικής στήριξης. Ο Έρικ Σοχάιμ, από τον ΟΣΑ, ε, πρόεδρος της ΝΤΑΚ, έχει ένα ε, κίνημα δημιουργήσει τους ε, φορολογικούς επιθεωρητές χωρίς σύνορα. Νομίζω ότι έχουμε αρκετή εμπειρογνωμοσύνη στα κράτη-μέλη και, και ίσως και μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, προωθήσουμε αυτή τη δημιουργία ικανοτήτων στέλνοντας ειδικού. Επίσης, τις πρωτοβουλίες διαφάνειας και αυτό πολύ σημαντικό. Κάποιες φορές Διερωτώ αν θα ήταν δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μια πρωτοβουλία και να διευρύνει το πεδίο των ε, πρωτοβουλειών ε, στις εξορρυκτικές βιομηχανίες, για παράδειγμα, να συμπεριληφθούν και οι ανανεώσιμες φυσικές πηγές ενέργειας. δεν μιλάμε μόνο για τα μεταλλεύματα, μιλάμε για την ε, δασοπονία, με παρανομιλοτόμηση, για του ε, λαθρο, τους λαθροκυνηγούς κτλ. Ε, πρέπει να κάνουμε πολλά λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά και τις παράνομες ώρες κεφαλαίων. Τώρα έχουμε το όλο θέμα της ανοιχτή βοήθειας, Open Aid, η DEFCO, νομίζω ότι έχει προχωρήσει. Αν δεν κάνω λάθος τουλάχιστον με αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Για παράδειγμα, πέραν της δημοσιοποίησης απλά ε, των στοιχείων για, το, για την βοήθεια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούσε να είναι, έχουμε ένα είδος κόκκινου κουμπιού. Κάτι που έκανε πρόσφατα η φιλανδική κυβέρνηση. Δηλαδή, πολύ απλά, με μια πολύ απλή τεχνική, οποιοδήποτε μπορεί να πληροφορεί για, μέχρι και για υπόνοιες ε, κατάχρησης ε, βοήθειας. Το ίδιο μπορεί να γίνει και από την πλευρά των ε, δικαιούχων, των αποδεκτών στις χώρες εταίρους. Να μιλήσω επίσης στις κρατικές επιχειρήσεις. Σε διάφορες χώρες αν υπάρχει αδιαφανής προεδρική διοίκηση ή κρατική διοίκηση, πολλές φορές γίνονται κάποια πράγματα με τους κρατικούς οργανισμούς, με τις κρατικές δομές, μέσα σε ένα στενό, κλειστό κύκλο σε αυτή τη δίκηση. Και νομίζω θα πρέπει να δούμε τι κάνει ο ΣΑ με τις ε, καλές ε, πρακτικές στον τομέα αυτών των κρατικών επιχειρήσεων. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει πιο πολύ τέτοιε πρωτοβουλίε. Τέλο. Για την ε, δυνατότητα του τύπου να ασκεί κριτική. Αυτό είναι σημαντικό για το Αζερμπαϊτζάν, που τα δεν είναι ακριβώ αναπτυσσόμενη χώρα, αλλά τέλο πάντων ένα από του πολιτικού κρατουμένου του Αζερμπαϊτζάν, συγκεκριμένα η κυρία Ισμαήλοβα, Χαντίτζα Ισμαήλοβα, κρατείται και έχει καταδικαστεί γιατί δημοσιοποίησε κάποιε πληροφορίε, κάποιε καταγγελίες ε, για τον πρόεδρο και την οικογένειά του, που τους εμπλέξει σε σκάνδαλο διαφθοράς. Και μιλάμε για την εταιρεία Τέλεια Σόνερα που δραστηριοποιείται και στη Φιλανδία, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Δεν πρέπει να είμαστε ούτε αφελεί ούτε τυφλοί, ούτε να δεχόμαστε προσωμιώσει μεταρρυθμίσεων. Αλλά πρέπει να είναι πραγματικέ μεταρρυθμίσει. Και αν θέλουμε, νομίζω ότι μπορούμε να τι ελέγξουμε αυτέ τι μεταρρυθμίσει που θέλουμε να προωθήσουμε για να μπορεί να ρέει ελεύθερα η βοήθειά μα για του αποδέκτε, του φτωχού για να προωθούμε τα δημόσια αγαθά. Ευχαριστώ, πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Πρόεδρος, η Κομισιόν μήπως θα θέλει το λόγο. Να μας πείτε και ποια είστε παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε και εμείς. Σούζαν Μπίρλαντα, επικεφαλής της Μονάδας Δημοσιονομικής Υποστήριξης στα πλαίσια του, της ΔΕΦΚΟ. Συνεργάζομαι δηλαδή και με άλλους συναδέλφους οι οποίοι ασχολούνται με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Θεωρούμε ότι εξαιτία της διαφθοράς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κονδυλίων που χάνεται στις αναπτυσσόμενες χώρες και συμφωνούμε ότι όλες οι χώρες χρειάζονται κάποιες εσωτερικές πολιτικές προκειμένου να έχουν βιώσιμη ανάπτυξη για το καλό των πολιτών τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ ενεργά υποστηρίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια χώρες και περιφέρειες προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια, η λογοδοσία και η επιτήρηση όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις και Αναφέρομαι στην πρωτοβουλία του Δεκεμβρίου του 2002 ένα σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και έχουμε και μια ανακοίνωση 2010 για την οικοδόμηση φορολογικών αποτελεσματικών υπηρεσιών στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα και να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής σε διεθνές επίπεδο και στα πλαίσια της συνδιάσκεψης στην Αντίσαμπέμπα ασχοληθήκαμε με το ζήτημα αυτό, θα ασχοληθούμε μάλλον με το ζήτημα αυτό. Θα παρουσιαστεί μια νέα φορολογική πρωτοβουλία προκειμένου να προωθηθούν φορολογικές μεταρρυθμίσεις από τις όμενες χώρες, επικεντρωνόμενος κυρίως σε φορολογικά ζητήματα διεθνών διαστάσεων. Θα ασχοληθούμε επίσης με την πρωτοβουλία της αύξησης των φορολογικών εσόδων και της καλύτερης δαπάνηση συνέχεια των εσόδων αυτών. Θέλουμε επίση να δημιουργήσουμε τι απαραίτητε υποδομέ για την καταπολέμηση τη διαφθορά και για τη στήριξη τη καταπολέμηση διαφθορά μέσω συγκεκριμένων πολιτικών και προγραμμάτων. Μεταρρύθμιση των φορολογικών υπηρεσιών, των οικονομικών υπηρεσιών, της καταπολέμηση της, των εγκληματικών δραστηριοτήτων και τη δημιουργία συγκεκριμένων υπηρεσιών για την καταπολέμηση της διαφθοράς μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης, ευαισθητοποίηση των πολιτών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών και των κοινοβουλίων. Συγκεκριμένα παραδείγματα μπορούμε να δώσουμε μέσω της εργαλειοθήκης που έχει προτείνει ο ΩΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο φοροδογικό τομέα, καθώς επίσης και στα μέσα τα οποία έχει προωθήσει η Transparency International τους στόχους ε, για την περίοδο μετά το 2015 όσον αφορά την παγκόσμια ανάπτυξη θέλουμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο προκειμένου να έχουμε εφαρμογή ενός νομοθετικού πλαισίου και την εφαρμογή εθνικών πολιτικών για τη μείωση της διαφθοράς. Στόχος 16, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος συνάδει με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς. Ο στόχος αυτός θα μπορέσει να αποτελέσει τη βάση για μια μελλοντική στρατηγική προσέγγιση. Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Θέλει να πάρει κάποιο άλλο το λόγο εξ ονόμου τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, πείτε μα και εσεί ποιος είστε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι ε, αναπληρωτής προϊστάμενος της μονάδας ε, που ασχολείται με την διαφθορά. Πρόκειται για την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αγώνα κατά της ε, διαφθοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ολοκληρωμένη προ πολιτική όσον αφορά την προαγωγή της ακεραιότητας και την αντιμετώπιση της διαφθοράς μέσω της νομοθεσίας. Είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεργασία επί του θέματος ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ε, κυρίως όσον αφορά ε, στην συνέχιση της έκθεσης ΚΡΙΜ και των σχετικών ψηφισμάτων. Εδώ υπάρχουν δύο σκέψεις που θέλω να αναφέρω για να ε, τοποθετηθώ στα σχόλια που έγιναν στην Επιτροπή. Καταρχάς να τοποθετηθώ στην εμπορική πολιτική και κατόπιν όσον αφορά τον προϋπολογισμό των κοινοτικών πόρων. Όσον αφορά λοιπόν την εμπορική πολιτική, σύσταση 55 του ψηφίσματος ΚΡΙΜ η σύσταση ε, έχει ως στόχο να συνδέσει την εμπορική πολιτική και τον αγώνα κατά της διαφθοράς. Μάλιστα η Επιτροπή συμφωνεί ότι ο αγώνας κατά της διαφθοράς είναι καθοριστική σημασίας ε, στις σχέσεις της με τις διάφορες χώρες. Η διαφθορά και κυρίως η δωροδοκία από το εξωτερικό αφορά τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις για να υπάρχουν ίσοι όροι για όλους. Οι εταίροι πρέπει να εφαρμόζουν τα ίδια στάνταρ τις προγραφές κατά της διαφθοράς. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει ήδη αυξήσει τη διαφάνεια ε, στους ε, δημόσιους διαγωνισμούς και στις σχέσεις με τους πελάτες. Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα για τις αναπτυσσόμενες χώρες και αυτά αφορούν τις προτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις γενικευμένες προτιμήσεις. Αυτό που ενδιαφέρει είναι επίσης η καλή διακυβέρνηση συμπεριλαμβανομένης και της ΟΝΚΑΚ, άρα δηλαδή υπάρχει σαφή διασύνδεση ε, όσον αφορά το σεβασμό των ε, ε, διεθνών συνθήκων για την αντιμετώπιση διαφοράς και αυτά σε σχέση με τις γενικευμένες προτιμήσεις. Οι συνάδελφοί μας ε, στην Γενική Διεύθυνση Εμπορίου αυτή τη στιγμή εργάζονται πάνω σε μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μελλοντική στρατηγική ε, που θα εγκριθεί αυτή η στρατηγική το φθινόπωρο. Στόχος είναι να διαπραγματευτούμε ειδικέ διατάξεις μελλοντικών εμπορικών συμβάσεων. Και η Επίτροπος Μάλμστρομ εχθές τόνισε αυτό το θέμα στην εισαγωγή της στην Επιτροπή Ίντα. Βεβαίως ε, θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω συζητήσεις για όλα αυτά κατά τους επόμενους μήνες. Ε, στοιχεία που έχουν σχέση με την εξωτερική πολιτική ε, και με την αντιμετώπιση της διαφθοράς αυτά τα στοιχεία ε, πρέπει να συνδυαστούν με τις γενικευμένες προτιμήσεις αλλά και ειδικέ ρήτρε για την αντιμετώπιση της αγοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτά αποτελούν ήδη ένα κομμάτι των συμφωνιών σύνδεσης. αλλά δηλαδή εδώ δεν πρόκειται μόνο για εμπορικές συμφωνίες και αυτό ισχύει για την τελευταία συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία. Αναφέρομαι στα άρθρα 3 και 14. Αυτά είναι ένα στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη και ως ένα πλαίσιο μετά το Κοτονού, τη συμφωνία του Κοτονού. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να στοχεύσουμε ε, στην Συμφωνία Κρίμ και συγκεκριμένα στη σύσταση υπαριθμών 19 που αφορά στον αποκλεισμό εταιριών που έχουν καταδικαστεί ως διεφθαρμένες και έχουν αποκλειστεί από τους διεθνείς διαγωνισμούς. Υπάρχει και μία νέα οδηγία για τους δημόσιους διαγωνισμούς και για τις παραχωρήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτείνει ένα σύστημα έγκαιρου εντοπισμού ε, με στόχο να προστατευτούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ε, οι τελευταίες, οι πρόσφατες εξελίξεις και εκεί επιτέχθηκε συμφωνία στις 29 Ιουνίου με στόχο να ακολουθήσει αργότερα μία νομοθετική πρωτοβουλία. Το 2016 θα έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις, οι ε, δημόσιοι διαγωνισμοί ε, θα είναι ασφαλείς από διαφθορά και αυτό είναι κάτι που ήθελα να υπογραμμίσω. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Οι ειδικοί έχουν το λόγο για να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο και να απαντήσω και στα ερωτήματα σε συντομία. Ευχαριστώ. Δύσκολα ε, μπορεί κανείς να συνοψίσει πολύ γρήγορα. Ε, όμως μπορώ ίσως να δώσω έμφαση σε κάποια από τα τελευταία σχόλια που ακούστηκαν και το λέμε και εμείς στην εκθεσή μας. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν έχουν κάποια αξιοζήλευτα χαρακτηριστικά που άλλοι δεν τα έχουν ε, Δηλαδή, εμπορικό θεματολόγιο μπορεί να συσχετιστεί με το αναπτυξιακό θεματολόγιο, το θεματολόγιο ασφάλειας κτλ. Δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος ε, παράγοντας αυτό αναπτυξιακής βοήθειας και αν καταφέρετε να έχετε μια καλύτερη κρατική προσέγγιση και συνεκτικότητα των πολιτικών στους τομείς αυτούς, αυτό είναι όφελος. Στην έκθεση λέμε ότι μιλάμε ακόμα για τις απαρχές αυτής της ε, συνεκτικότητας πολιτικής δεν έχει προχωρήσει ακόμη. Πρέπει επίσης να διδαχθείτε από ένα από τα πιο φιλόδοξα πειράματα, μπορούμε να τα πούμε έτσι, για την καταπολέμηση της διαφθοράς τα τελευταία χρόνια, με μεταρρυθμίσεις για το κύμα της διεύρυνσης. Δεν βλέπουμε ότι αυτό μπόρεσε να μεταφραστεί ε, και σε μέτρα καταπολέμησης διαφορά στην αναπτυξιακή βοήθεια. Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικές οι μένα τις δε χώρες, όμως θα μπορούσε να, υπάρξει, ε, να υπάρξουν κάποια διδάγματα. Τώρα, για τους δείκτες, για να δώσω κάποιες απαντήσεις. Ε, πολλές φορές μας τίθεται το ερώτημα για τους δείκτες και πώς μπορούμε να τα μετράμε καλύτερα αυτά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν χρησιμοποιούν κάποια από τα γνωστά ε, μέτρα που δίνει η Transparency International, Παγκόσμιος Τράπεζα κτλ. Από τη στιγμή που δεχτούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένα και μόνος δείκτης για πολλά διαφορετικά επίπεδα διαφθορά. θα πρέπει δηλαδή να αρχίσουμε να διευκρινίζουμε τους τομείς που θέλουμε να μετρήσουμε, το είδος της διαφθοράς, τα αποτελέσματα και τα προγράμματα. Μετά πάμε σε συγκεκριμένους τομείς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα εργαλεία όπως είναι οι περιφερειακές παράμετροι ή πιο από ομαδοποιημένα στοιχεία που δίνουν μια πιο καλή βάση για τον ετομισμό των μεταρρυθμίσεων και των επιπέδων διαφθοράς σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική στήριξη και την αρισιμότητα. Πολλά ακούστηκαν σχετικά. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει αυτή την ε, αρχή της αεροεσιμότητας για την κακή διαχείριση των ε, κονδυλίων. Βλέπουμε στο πρόγραμμα γειτονία έχουμε την αρχή περισσότερα για περισσότερα, more for more. Δεν βλέπουμε να γίνεται με τον ίδιο τρόπο αυτή ε, η προσέγγιση να ακολουθείται και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τέλος. το ότι θέλετε να εφαρμόσετε την αρεσιμότητα δεν αποτελεί από μόνο του μια στρατηγική. Υπάρχουν και το ακούσαμε πολλά διαφορετικά είδη στήριξης, αλλά δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία συμφωνία για το αν δουλεύει, πόσο δουλεύει το κάθε σύστημα. Επομένως, πρέπει ίσως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να να δει τα πράγματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ω αναπτυξιακό παράγοντα και να δώσει επιχειρησιακή καθοδήγηση στο προσωπικό και στι αντιπροσωπείς της Ένωσης ανά τον κόσμο. Αυτό ήταν χρήσιμο, να του δώσει οδηγίε. Να συνεχίσω κι εγώ πώς μπορούμε να συνδυάσουμε διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά την αιρεσιμότητα και πιο συγκεκριμένα τι μπορούμε να κάνουμε σε χώρες όπου έχουμε παρόντες και άλλους παράγοντες λιγότερο αυστηρούς όσον αφορά την αιρεσιμότητα. Κοιτάξτε, όντως στην πράξη βλέπουμε ότι υπάρχει μια χώρα στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών όπου υπάρχουν πολλές χώρες δωρητές που έχουν επέμβει προκειμένου να αντιμετωπίσουν ένα σκάνδαλο διαφθοράς. Σε έναν από τους τομείς της οικονομίας υπήρχε ένα σημαντικό σκάνδαλο διαφθοράς και οι δωρητές είπαν ότι θα αποσύρανε τότε την χρηματοδότησή τους. Η κυβέρνηση είπε πόσα χρήματα θα μας πάρετε προκειμένου να πάμε σε άλλους δωρητές και να τους ζητήσουμε τα χρήματα αυτά και να αντισταθμίσουμε τα χρήματα που θα μας πάρετε. Όταν όμως συνειδητοποίησαν ότι θα επηρεαζόταν από το σκάνδαλο αυτό και η βαθμολόγηση του οίκου αξιολόγηση Moody's και ότι αυτό με τη σειρά του θα επηρέαζε το βαθμό επενδύσεων στη χώρα αυτή, τότε άλλαξαν στάση και υιοθέτησαν μια διαφορετική, πιο προσεκτική προσέγγιση. Νομίζω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να ασκήσουμε πίεση μέσω συγκεκριμένων νομισμάτων ή εθνικών προσεγγίσεων σε κάποιες χώρες. Είναι περισσότερο το να προσπαθήσει να αντιράσει κανείς τη φήμη μιας χώρας, αυτό το οποίο μπορεί να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά. Θα ήθελα να αφαιρθώ τώρα στο ζήτημα αυτό της υποκρισίας που θίξατε, ότι θα περιμένουμε πολλές φορές από αναπτυσσόμενες χώρες να φτάσουν το επίπεδο διαφάνειας που έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι και στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς. Για ποιο λοιπόν να θεωρούμε ότι οποιοδήποτε ευρώ πηγαίνει σε μία αναπτυσσόμενη χώρα ενδεχομένως να αποτελέσει αντικείμενο διαφθορά, στη στιγμή που κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί ακόμα και σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Ενδεχομένως λοιπόν θα πρέπει να δούμε το εξή και ξέρω ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πει κανεί. Ποιο βαθμό διαφθοράς μπορούμε να αποδεχθούμε όταν συγκρίνουμε την κατάσταση σε μια αναπτυσσόμενη χώρα με τους στόχους ανάπτυξης που έχουμε για τη χώρα αυτή, νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και τους δυο σας και όλους σας βασικά σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων που είχαμε. Δεν έχουμε συγκεκριμένη προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για αυτή τη γνωμοδότηση γιατί η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, η ΛΥΜΠΕ, δεν μας έχει επιβεβαιώσει ακόμα το δικό της το χρονοδιάγραμμα. Συνεχίζουμε λοιπόν και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης «Ανθρωπιστική κρίση στο Νότιο Σουδάν». Ιδιαίτερα επίκαιρο το ζήτημα. Έχουμε την τέταρτη επέτειο από την ανεξαρτησία του Νοτιού Σουδάν Συνεχίζεται όμως η βία με αποτέλεσμα 2 εκατομμύρια άνθρωποι να έχουν εκτοπιστεί. 500 περίπου χιλιάδες κάτοικοι της νο... του Νότιου Σουδάν, κυρίως παιδιά, έχουν πάει σε γειτονικέ χώρες. Περίπου 2,75 εκατομμύρια άνθρωποι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Εθνή, δηλαδή το 1 τέταρτο περίπου του πληθυσμού, θα πλήγονται μέχρι το τέλος του έτους από επιστηστική ανασφάλεια. Μολονότι λοιπόν εμβαθύνονται και συνεχίζονται τα προβλήματα, η συνεχιζόμενη βία έχει θέσει εν κινδύνο και την ίδια την παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Και βέβαια εμείς ως Επιτροπή Ανάπτυξη ανησυχούμε ιδιαίτερα για την κατάσταση των ανθρώπων στη χώρα αυτή. Θα μπορούσαν ε, οι ομιλητές μας να έρθουν εδώ πέρα και να πάρουν επίσης και τις καρτέλες τους μαζί τους. Συγγνώμη, προχώρησα πολύ γρήγορα, λέει ο Πρόεδρος. Well, now we Λοιπόν, τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε πάλι. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε ανάμεσά μας ε, τους εκλεκτούς μας ε, ομιλητές ε, για το ζήτημα αυτό. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ζαν Λουί Ντεμπρόερ από την DG ECO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Τσόις Λούμα από το Παγκόσμιο Επιστηστικό Πρόγραμμα, την κυρία Λάιλα Πιέτερς η οποία εργάζεται για τη UNICEF, καθώς επίσης και τον κύριο Όσκαρ Μούντια από το UNHCR των Ηνωμένων Εθνών. Ο πρώτος ομιλητής ήταν ο κύριος Δεμπρόερ. Σας παρακαλώ πολύ, μιλήστε το πολύ 5 με 7 λεπτά. Ξέρω ότι δεν το δίνω πάρα πολύ χρόνο, αλλά ελπίζω να τα καταφέρετε. Έχετε το λόγο. Γεια σας. Κυρίε και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, 14 Ιουλίου σήμερα. Αν με επιτρέπετε να μιλήσω γαλλικά λοιπόν, καθώ τεχνική εορτή για τη Γαλλία. Βέβαια είτε στα αγγλικά είτε στα γαλλικά. Αυτό που έχω να πω φοβούμε είναι η άκρος ανησυχητική δεινή ανθρωπιστική κατάσταση. Όπως είπατε λοιπόν και εσείς στην εισαγωγή σας, ε, κύριε Πρόεδρε, συνεχίζει τα γαλλικά Ομιλητή, ε, η κρίση στο Νότιο Σουδάν, που είναι σε επίπεδο 3 στην ιεράρχηση του Ηνωμένου το του τη ομοθεσία της κρίση, είναι η μεγαλύτερη, σοβαρότερη ανθρωπιστική κρίση σήμερα στον πλανήτη. Περίπου 1,6 εκατομμύρια εκτοπιστέντες, εσωτερικά εκτοπιστέντες, 600.000 πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες, και 165.000 ε, στις ζώνες προστασίας αμάχων που είναι κοντά στις βάσεις ε, των ΗΕ. Θα επανέλθω σε αυτά τα στοιχεία. Απλά θέλω να επιμείνω ε, ευθύς εξ στον όλο και πιο περιφερειακό χαρακτήρα της κρίσης λόγω του αποσταθεροποιητικού αντικτύπου ε, που έχει και η μετακίνηση των ε, πληθυσμών προσφύγων και εξωτερικά εκτοπιστέντες. Ο κύριος Στυλιανίδης, Χρήστος Στυλιανίδης, ε, Επίτροπος Αρμόδιος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια, πριν από έξι εβδομάδες μετέβη στο Νότιο Σουδάν, πέρασε και από την Αιθιοπία και έδωσε σαφή μηνύματα. Τα επανέλαβε εν συνεχεία και μέσω της κοινή ανακοίνωσης τύπου με την είπατε εκπρόσωπο κυρία Μογκερίνη. Τα μηνύματα αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι μηνύματα αλληλεγγύης απέναντι ε, στο λαό του Νότιου Σουδάν που χυμάζεται και είναι απογοητευμένος, απελπισμένο. Αναγνώριση και στήριξη που πρέπει να δοθεί στα ανθρωπιστικά συνεργεία που πρέπει να εργαστούν υπό άκρος απαιτητικές συνθήκες. Να έχουμε υπόψη επίσης ότι από το Δεκέμβριο του 2013 30 εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας έχασαν τη ζωή τους ε, στο Νότιο Σουδάν και ότι οι βάσεις, οι αποθήκες 10 τροπιστικών οργανώσεων ε, λαιλατήθηκαν ή καταστράφηκαν από τον ε, Απρίλιο και μετά. Με αυτά τα στοιχεία νομίζω ε, έχετε έτσι μια εικόνα για το πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες εργασίας για τους ε, εργαζόμενους στο ανθρωπιστικό ε, τομέα. Ο κύριος Τηλιανίδης επίσης τόνισε ότι η κατάσταση είναι αδύνατον, είναι αφόρητη και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αφόρητη υπό δύο ενείς, σε δύο άξονες. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τα πολιτικά αίτια έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανθρωπιστικές επιπτώσεις της σύγκρουσης. Δύο ανδρών ουσιαστικά ή δύο φατριών που αγωνίζονται για την εξουσία και τα προνόμια της εξουσίας και που περιφρονούν όσο πιο ε, απόλυτα γίνεται την οδύνη που μπορεί αυτή η αντιπαλότητα να δημιουργεί στο λαό για τον οποίο είναι ή ήταν υπεύθυνοι και για την προστασία του βέβαια. Θύμισε, λοιπόν ο κύριος Στυλιανίδης και στα μέλη της κυβέρνησης αλλά και στους ηγέτες αντιπολίτευσης με τους οποίους συναντήθηκε τις ευθύνε που έχουν. Επίσης, η κατάσταση είναι αφόρητη και σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες που ζητούνται από τη διεθνή ανθρωπιστική κοινότητα. Οι συνάδελφοι και συνεισηγητές ε, σήμερα θα σας ε, εξηγήσουν ε, τη σημασία, το πόσο σημαντικές είναι οι ανάγκες. Όλο και πιο δύσκολο καθίσταται οι χρηματοδότες να μπορούν να ανταποκριθούν στα αιτήματα και στις προσδοκίες, Λάμβοντας υπόψη και ένα πολύ γνωστό στην Επιτροπή σας φαινόμενο, κύριε Πρόεδρε, η τί τον πολλαπλασιασμό των ανθρωπιστικών κρίσεων μεγάλης εμβέλειας ε, είναι άνευ προηγουμένο πολλαπλασιασμό των κρίσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Άμα την επιστροφή του κύριο Στυλιανίδης ε, συμπροείδρευσε ε, στις 16 Ιουνίου με τον κύριο Ομπράιεν, τον νέο υπεύθυνο, στη Γενέβη, ε, τη δεύτερη επιχείρηση συλλογής πόρων μετά από αυτή που έγινε το Μάρτιο στην περιοχή. Πράγματι συγκεντρώθηκαν πόροι και ε, σημειώθηκαν δεσμεύσεις ε, για δωρεές συνολικού ύψους 245 εκατομμυρίων. Δεν είναι αμεληταίο το ποσό, αλλά γνωρίζουμε ήδη ότι είναι ανεπαρκές για να καλύψει τι ανάγκε όπως τι υπολογίζουμε μέχρι τα τέλη του έτου. Σε ένα τελευταίο σημείο, το οποίο θα ήθελα να επιμείνω κύριε Πρόεδρε, πριν δώσω το λόγο στου συναδέλφου μου. Πρόκειται για την εξαιρετική βία η οποία σημαδεύει την αντιπαράθεση αυτή. Θα διαβάσω ένα κείμενο, σύντομο κείμενο, στα αγγλικά. Τουλάχιστον 172 γυναίκες και κορίτσια έχουν απαχθεί και άλλες 79 υποβλήθηκαν, ε, υπέστησαν ε, ε, κακοποίηση και βιασμό, ομαδικό βιασμό. Μάλιστα υπήρξαν και θάνατοι πάνω ε, από πέντε χωριά ε, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν ε, μετά από μαδικό βιασμό γυναίκες και κορίτσια. Πρόκειται για το απόσπασμα μια έκθεση της Amnesty International Flash Human Rights 29 Ιουνίου δημοσιεύτηκε με μαρτυρίες από επιζώντες της αρνητικής επίθεσης ε, που ε, εξαπέλυσε η κυβέρνηση. Το Συμβούλιο Ασφαλείας υιοθέτησε ένα ψήφισμα τον Ιούνιο και ξεκάθαρα αναφέρεται σε εγκλήματα πολέμου. Λέει ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστέψει κανείς ότι έχουμε ε, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν και από την κυβέρνηση και από τις αρχές αντιπολίτευσης και το ίδιο ψήφισμα μιλά και ξεκάθαρα για δείγματα περαιτέρω εθνικοποίησης της αντιπαράθεσης. Τι βλέπουμε στον ορίζοντα. Μπορεί να πούν και άλλοι βέβαια. Ήρθατε να λέμε ότι είναι ανθρωπιστική η, λύση, αλλά, η κρίση, αλλά η λύση είναι πολιτική. Δεν βλέπουμε όμως να διαφέρονται λύσεις πρόθεσμα και σε αυτό έρχεται να προσθεθεί και η, η θεαματική επιδείνωση ε, της οικονομίας στο Νότιο Σουδάν. Μια χώρα που βρίσκεται στο χείλος της χρεοκοπίας λόγω της σύγκρουσης αυτής, της αντιπάρτησης αυτής. Εδώ θα σταματήσω εγώ κύριε Πρόεδρε, αφού πρώτα ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που έλαβε την πρωτοβουλία να μας καλέσει εδώ σήμερα είναι μια κρίση που δεν μπορούμε να λησμονούμε γιατί έχουμε ηθική ανθρωπιστική ευθύνη ε, και αυτή η κρίση του Νότιου Σουδάν είναι η κατεξοχήν κρίση που δεν μπορούμε να λησμονήσουμε. Ευχαριστώ. Uh, Εμεί ευχαριστούμε. Η κυρία Λούμα είναι επόμενο ομιλητής. παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Το Νότιο Σουδάν ε, αντιμετωπίζει τα σημαντικότερα επίπεδα επιστηστικής ανασφάλειας από την ανεξαρτησία του. Να 40%, 4,6 εκατομμύρια άνθρωποι δηλαδή, θα αντιμετωπίσουν τις επόμενους τρεις μήνες απόλυτη πείνα. Πάρα πολλά παιδιά κάτω της ηλικία των 5 ετών λιμοκτονούν. Πέντε από τις 10 περιφέρειες της χώρας αντιμετωπίζουν πολύ ψηλά επίπεδα επιστημικής ανάσφειας. Πιέζεται πάρα πολύ η οικονομία της χώρας, καθότι μειώνονται τα έσοδα και υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές αμυντικές δαπάνες. Η τιμή των καυσίμων, αυξάνεται όλο και περισσότερο, δεν υπάρχουν τα απαραίτητα προϊόντα και αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ τον τοπικό πληθυσμό και ιδίω στους πιο φτωχούς. Η κλιμάκωση αυτή της βίας που έχουμε δει πρόσφατα σε ορισμένα κρατήδια της χώρας αυτής οξύνει ακόμα περισσότερο την επιστημική ανασφάλεια. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ατόμων που έχουν εκτοπιστεί. Πάρα πολλοί έχουν πάει στα κέντρα των ΗΕ Εθνών ζητώντας προστασία. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες των οποίων έχει καταστραφεί η ζωή ή το βιός τους. Η κρίση αυτή συμβαίνει κάτι διάρκεια της περίοδου της σποράς, πραγματοποιήσουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν θα καταφέρουν να σπείρουν τα χωράφια τους και αυτό θα εντείνει περισσότερο την επιστημική κρίση. Λαμβάνοντας λοιπόν όλα αυτά υπόψη μας, εμείς ως παγκόσμιο πρόγραμμα επισητισμού προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον πληθυσμό της χώρας στις περιοχές που πλήττονται από, την, από τη διένεξη αυτή προσπαθήσαμε ήδη από τα αρχές του 2014 να κινήσουμε το μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης και δράσης. Δόθηκε λοιπόν, δόθηκαν τα παρέτα τρόφιμα στους ανθρώπους που πλήττονται στις περιοχές αυτές. Προσπαθήσαμε να δώσουμε διαέρος τα παρέτα προϊόντα. Το WFP και οι εταίροι τους έχουμε 27 κινητές μονάδες που βοήθησαν τον πληθυσμό σε 90 περίπου περιοχές της χώρας. Οι επιπτώσεις όμως της ε, χώρας δεν ε, οι επιπτώσει αυτές δεν πλήττουν μόνο το βόρειο τμήμα της χώρας. Βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και λιγότερες ε, παρεχόμενες υπηρεσίες που οδηγούν σε επιστηστική ανασφάλεια ακόμα και σε περιοχές οι οποίες ήταν μέχρι πρόσφατα πιο σταθερές. Προσπαθούμε εμείς ως παγκόσμιο επιστηστικό πρόγραμμα να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αυξήσουμε την ανθεκτικότητά του και να οδηγήσουμε σε μια κάποια ευημερία. Έχουμε λοιπόν ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2014 προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την επιστηστική κρίση στη χώρα. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε τον πληθυσμό όσον αφορά την πρόληψη και όσον αφορά την αντιμετώπιση της, των πληθυσμών εκείνων που πλήττονται από την επιστημική ανασφάλεια. Προσπαθούμε να δώσουμε δελτία προκειμένου να μπορούν οι άνθρωποι να αγοράζουν κάποια τρόφιμα. Μέσω όλων αυτών των προσπαθειών καταφέραμε να βοηθήσουμε 2,2 εκατομμύρια άτομα το 2014. Η γενικότερη υποστήριξη που δόθηκε από τους ανθρωπιστικούς μας εταίρους και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας βοήθησε πάρα πολύ και θα θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας. Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε ένα πολύ αντίξω περιβάλλον το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή έχει κλιμακωθεί η βία σε πάρα πολλέ περιοχέ τη χώρα δεν μα επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση στι πιο ευάλωτε ομάδε του πληθυσμού, ιδίω στι πιο δύσκολε, δύσβατε περιοχέ που πλήττονται από τι διενέξει. Πολλέ φορέ δεν έχουμε πρόσβαση στον πληθυσμό αυτό ή άλλε φορέ ενώ επιτρέπεται η πρόσβαση είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για κάποιε ανθρωπιστικέ ομάδε να φτάσουν σε αυτέ τι περιοχέ. Η WFP λοιπόν μείωσε τις κινητές ομάδες στις περιοχές αυτές προκειμένου να προστατεύσει τους ανθρώπους που εργάζονται για την προστασία του πληθυσμού. Οι ίδιες οι κοινότητες πολλές φορές των επιτόπου κατοίκων μας λένε ότι δεν πρέπει να πάμε στις περιοχές αυτές γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είμαστε σε επαφή με τη διεθνή ανθρωπιστική κοινότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε καταφέρει να δώσουμε κάποια κοιτή επιβίωσης που ε, περιλαμβάνουν σπόρους, βασικά τρόφιμα, ε, εντομοποθητικά ε, μπισκότα και άλλα τέτοια βασικά προϊόντα. Τα δώσαμε αυτά σε κάποιες περιοχές στις οποίες δεν μπορούμε να μείνουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ανασφάλεια επεκτείνεται τώρα σε κάποιες περιοχές που στο παρελθόν ήταν σταθερές. Η μεταφορά λοιπόν βασικών προϊόντων στα πλαίσια του Νοτιού Σουδάν έχει καταστεί ακόμα πιο δύσκολη. Δεν υπάρχουν πλέον ασφαλείς διάδρομοι προκειμένου να καταφέρουμε να διοχετεύουμε βασικά προϊόντα σε όλες τις περιοχές της χώρας. Επίσης είδαμε πολλά φαινόμενα λαιλασίας, κυρίως φορτηγών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια και κάποια βασικά προϊόντα. Και ως αποτέλεσμα χρειάστηκε να αναστείλουμε προσωρινά τη μεταφορά των βασικών αυτών προϊόντων, κυρίως στους δυτικούς διαδρόμους. Η μεταφορά επίσης των τροφίμων στους διαδρόμους αυτούς γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη καθότι θα πρέπει τα φορτηγά αυτά να περνάνε από κάποιες περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο διαφόρων ένοπλων δυνάμεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε εμεί να διοχετεύσουμε τη βοήθεια αυτή σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εντελώ κατακαιρματισμένο. Χρησιμοποιούμε την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών, την UNMIS, προκειμένου να καταφέρουμε να παράσχουμε βασικά προϊόντα σε κάποιες επικίνδυνες περιοχές. Κάθε χρόνο ένα 60% της χώρας ε, δεν ε, είναι προσβάσιμο κυρίως λόγω των πλημμύρων, όταν ξεκινάει δηλαδή η περίοδος των προχοπτώσεων. Στις περιόδους λοιπόν αυτές μειώνεται πάρα πολύ η έκταση κατά την οποία μπορούν να ταξιδέψουν ε, όλα αυτά τα φορτηγά τα οποία μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και βασικά προϊόντα. Εμείς δεν καταφέραμε εξαιτία λοιπόν των κλιματικών αυτών συνθηκών αλλά και εξαιτία ε, των ε, διενέξεων και των τοπικών συγκρούσεων να δώσουμε και να παράσχουμε όλη την απαραίτητη ε, ανθρωπιστική βοήθεια. ότι θέλουμε να μειώσουμε το κόστος των δράσεών μας αυτών, θα χρειαστούν παρόλα αυτά παραδόσεις μέσω αεροπλάνων σε ορισμένες περιοχές. Αυτό αποτελεί μια ίστατη λύση προκειμένου να καταφέρουμε να φτάσουμε στους πιο απομονωμένους πληθυσμούς. Το 2015 είχαμε κάποιες περικοπές όσον αφορά τους πόρους μας. Χρειάστηκε λοιπόν να επικεντρωθούμε περισσότερο σε κάποιους πληθυσμούς που πλήττονται περισσότερο και να κάνουμε μια ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Έγιναν λοιπόν κάποιες περικοπές, δεν καταφέρνουμε πλέον να καλύψουμε περίπου 250.000 πρόσφυγες και χρειάστηκε να επικεντρωθούμε κυρίως στις περιοχές εκείνες που πλούνται περισσότερο εξαιτία των διενέξεων. Μολονότι υπάρχουν κάποιοι πληθυσμοί επιτόπου που περνοσμένα χρειάζονται τρόφιμα, παρόλα αυτά εμείς καταφέραμε να παρέχουμε βοήθεια κάθε δύο ή τρεις μήνες, ενώ στο παρελθόν η συμβολή μας συνέβαινε σε μηνιαία βάση. Χρειάζεται λοιπόν να καταφέρουμε να καλύψουμε το δημοσιονομικό αυτό κενό. 180 εκατομμύρια ευρώ χρειαζόμαστε τους επόμενους έξι μήνες. Αν δεν έχουμε τους απαραίτητους αυτούς πόρους θα χρειαστεί να κάνουμε περαιτέρω περικοπές και περαιτέρω ιεράρχηση προτεραιοτήτων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού τα οποία χρειάζονται περνοσμένα τρόφιμα και παρόλα αυτά δεν θα έχουν πρόσβαση την ανθρωπιστική επιστηστική αυτή βοήθεια. Μολονότι γίνεται προσπάθεια από τη διεθνή κοινότητα για να επιληθεί η τοπική κρίση, οι πολίτες χρειάζονται απεγνωσμένα ανθρωπιστική και επιστηστική βοήθεια και εμείς ως παγκόσμιο επιστηστικό πρόγραμμα θα συνεχίζουμε να παρέχουμε βοήθεια στους ανθρώπους αυτούς. Ευτυχώς είχαμε την βοήθεια την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε για τη δημοσιονομική σα υποστήριξη, αλλά και την επιτόπου βοήθεια που μα παρήσχατε, προκειμένου πραγματικά τα προϊόντα αυτά και τα τρόφιμα αυτά να φτάσουν του τελικού αποδέκτε. Σα ευχαριστώ. Επόμενος μιλητής, ε, η κυρία Πίτερ. Καλησπέρα σας. Ε, σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι από την ε, ε, Ευρωπαϊκή, Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Δράσης, από την ΔΕΦΚΟ, από την ΕΦΚΟ, του συναδέλφους, από τα Ηνωμένα Έθνη και από την Κοινωνία των Πολιτών δεν θα χρησιμοποιήσω το PowerPoint γιατί δεν έχουμε χρόνο και θα πέρασω κατευθείαν στο θέμα μου. Καταρχάς ε, να σου πω ότι μιλώ εκ μέρους της ε, UNICEF του Νότιου Σουντάν αλλά και εκ μέρους της UNICEF και θέλω να εκφράσω τις ευχαριστήσεις μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως στην Γενική Διεύθυνση DEFCO για την πολύ γενναιόδορη υποστήριξή της ε, κατά τα τελευταία χρόνια. Λάβαμε 15 εκατομμύρια ευρώ από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Και με αυτήν την οικονομική υποστήριξη μπορέσαμε να κατορθώσουμε πάρα πολλά, σώσαμε πολλές ζωές, παιδιών επίσης. Να σας πω, λοιπόν, με αυτή την υποστήριξη από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ αλλά και από άλλα κρατημέλη μπορέσαμε να σώσουμε τη ζωή 63.000 παιδιών από υποσυτισμό μπορέσαμε να εμβολιάσουμε πάνω από 6 εκατομμύρια παιδιά, με το εμβόλιο της πολιομελίτητας επανήλθαν αυτά στο σχολείο. Πολύ σημαντικά όλα αυτά λόγω της γενναιόδορης υποστήριξης. Παρ' όλα αυτά το μέλλον των παιδιών στο Νότιο Σουδάν είναι ιδιαίτερα ζωφερό. Πριν από λίγες ημέρες ε, μπορέσαμε να γιορτάσουμε την τέταρτη ημέρα ανεξαρτησίας του Νότιου Σουδάν. Ε, σε αυτές, αυτά τα τέσσερα χρόνια υπήρξαν ε, μα πραγματικά κατάφορες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών. Μιλάμε για δολοφονίες. Η δολοφονία παιδιών, γυναικών, κοριτσιών πρέπει να σταματήσει. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η διεθνή κοινότητα να δραστηριοποιηθεί έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το, αυτή η ομίδια η διεθνής κοινότητα οφείλει να κινητοποιηθεί, να ενώσει τις δυνάμεις της για να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση έτσι ώστε σε πρώτη φάση να μπορούμε να μετρήσουμε αυτές τις παραβιάσεις αλλά και να προσφέρουμε βασικές υπηρεσίες. Όπως είπε και ο συνάδελφός μου από το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισητισμού ε, χρειαζόμαστε χρήματα ε, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ανακαλύψουμε ε, νέους τρόπους χρηματοδότησης Βλέποντας λοιπόν τη χρηματοδότηση στις αναπτυσσόμενες χώρες, εκεί έχουμε περισσότερα κονδύλια. Πρέπει να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις πράξεις μας και τις δραστηριότητές μας. Και έχουμε να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις θα θέλαμε να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα προγράμματα ε, επισητισμού Αυτά τα οργανώνουμε σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Ψητισμού αλλά και με διεθνείς εταίρους. Να προσπαθήσουμε τα παιδιά να επανέλθουν στο σχολείο και να δούμε πώς το πρόγραμμα ειρήνης που έχει χρηματοδοτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς αυτό μπορεί και αυτό να συνεχιστεί. Και εδώ θα ήθελα να σταματήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία, δεν χρησιμοποίησατε όλο το χρόνο που σας είχε ε, διατεθεί. Ο κύριος Μούντι είναι ο τελευταίος ομιλητής. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη δυνατότητα που μας δώσατε να σας μιλήσουμε. Η δική μου δουλειά είναι πολύ απλή. Μετά τους τρεις προλαλήσαντες, ε, τα περισσότερα έχουν υποθεί. Εγώ απλά θα αναφερθώ στην περιφερειακή διάσταση της κρίσης. Γιατί Νομίζω σήμερα το απόγευμα θίξαμε κυρίως την εσωτερική διάσταση της κρίσης, αλλά υπάρχει και ένα περιφερειακό στοιχείο. Ε, θα σας κάνω μία ε, παρουσίαση με PowerPoint, γιατί αυτή η παρουσίαση αφορά και τις τέσσερις χώρες που έχει πλήξει η κρίση. Να πω λοιπόν καταρχήν, πριν από δέκα χρόνια και ένα μήνα, όταν υπογράφηκε η συμφωνία είχαμε πολύ λιγότερους ε, πρόσφυγες Σουδανέζους. Τώρα έχουμε 738.000 πρόσφυγες από τον Νότιο Σουδάν σε διάφορες χώρες της περιοχής. Πρόσφατα εντάθηκαν οι συγκρούσεις, οι ένοπλες συγκρούσεις στο Απανέλ και αυτό οδήγησε όχι μόνο σε εσωτερικό εκτοπισμό στο νότιο Σουδάν, αλλά και στο ίδιο το Σουδάν. Βλέπουμε ότι το προφίλ των προσφύγων στην περιοχή είναι κυρίως γυναίκες και παιδιά. Το 80% των προσφύγων είναι γυναίκες και παιδιά. Μιλάμε για πολύ, μια πολύ ευάλωτη ομάδα. Ως εκ τούτου η δραστηριότητά μας πρέπει να είναι προσαρμοσμένη σε αυτό το προφίλ. Στο Νότιο Σουδάν, ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ε, πρόσφυγες, Σουδανέζους πρόσφυγες, η πλειοψηφία αυτών είναι στο Απανέλ που είναι, όπως ακούσατε από τους προλαλήσαντες, το ε, επίκεντρο των ε, ένοπλων συγκρούσεων. Αυτούς πρέπει να τους προστατεύσουμε και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση να προσφέρουμε υλική βοήθεια σε μια περιοχή όπου υπάρχουν ε, αυτές οι συγκρούσεις. Αυτό είναι ακριβό και σχεδόν και αδύνατο. Κατόπιν τούτου, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, αυτή είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, αλλά πρέπει να την κάνουμε διότι διακυβεύεται η ζωή ανθρώπων. Δεν θα μιλήσω για τους αριθμούς που βλέπετε εκεί, απλά πολύ σύντομα να πω ότι τα, βιβλία που, τα στοιχεία που βλέπετε πάνω δεξιά είναι ο αριθμός των προσφύγων που περιμένουμε να ε, έρθει από τον Νότιο Σουντάν μέχρι το τέλος του έτους. Μέσα στο ίδιο το Σουντάν βλέπετε ότι έχουμε περίπου 5.000 λιγότερους από τους ε, προβλεπόμενους και αυτό σας δείχνει τη δραματική κατάσταση που προκύπτει. Στην επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Και αυτή η διαφάνεια είναι απεικόνηση του μεγέθους της, του εκτοπισμού τόσο εσωτερικά μέσα στο Νότιο Σουδάν όσο και εξωτερικά. Μιλάμε λοιπόν συνολικά για 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν πληγεί, εσωτερικά εκτοπισμένοι 1,5 ε, εκατομμύρια, ε, στο Νότιο Σουντάν 650.000 και βέβαια και στις ε, διάφορες χώρες, θα σας αναφέρω αργότερα. Εδώ τώρα, επόμενη διαφάνεια. Εδώ, όπως είπε και ο κύριος Δεμπρός, βλέπουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει πολιτική λύση. Γιατί η ανθρωπιστική βοήθεια είναι κακή βοήθεια η πολιτική λύση είναι το βασικό. Και γι' αυτό κάνουμε έκκληση να υπάρξει πολιτική λύση για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Δεν θα αναφερθώ στα μεμονωμένα στοιχεία που αναφέρονται στη διαφάνεια. Θα ήθελα μόνο να υπογραμμίσω ότι στο Νότιο Σουδάν έχουμε δυσκολία να προστατεύσουμε τους ε, πρόσφυγες. Επόμενη ε, διαφάνεια παρακαλώ. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι το εξής. Υπάρχει η ανάγκη να στηρίξουμε και τις περιοχές που πάνε εκεί οι πρόσφυγες. Στο βόρειο κομμάτι της Ουγκάντα, της Κένιας, στο ανατολικό κομμάτι της Κένιας, στο νότιο κομμάτι του Σουντάν. Δηλαδή οι πρόσφυγες πάνε ε, σε περιοχές όπου ήδη υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Άρα δηλαδή και αυτές οι περιοχές δεν μπορούν εύκολα να φιλοξενήσουν τους πρόσφυγες. Όσοι βρισκόμαστε σε αυτόν τον τομέα ξέρουμε ότι εκεί καταρχήν πρέπει να προσφερθεί η βοήθεια. Γιατί βέβαια αν δεν υπάρχει ειρήνη σε αυτές τις περιοχές δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους ε, πρόσφυγες καλούμε τις κυβερνήσεις που πλήττονται να στηριχτούν έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη προστασία. Πρέπει να πω ότι οι κυβερνήσεις και των τεσσάρων κρατών έχουν ανοίξει ε, τα σύνορά τους ανοιχτά και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί το πρώτο βέβαια βήμα για να προστατεύσει πρόσφυγες είναι να είναι ανοιχτά τα σύνορα. Αυτές λοιπόν οι χώρες έχουν κρατήσει ανοιχτά τα σύνορα και έχουν προσφέρει ε, γη, υπάρχει τέτοια δυνατότητα περισσότερες χώρες. Έχουμε λοιπόν αρκετή γη για να τους φιλοξενήσουμε και όπου δεν υπάρχει αυτή η γη δεν είναι λόγω έλλειψης βούλησης αλλά διότι υπάρχει διαμάχη ανάμεσα στην κεντρική και την περιφερική κυβέρνηση και αυτά πρέπει να επιληθούν πριν προσφερθεί η απαραίτητη έκταση για τους πρόσφυγες. Και στις τέσσερις χώρες έχουμε καταβλισμούς ε, και θα σας δείξω και τα απαραίτητα στοιχεία αργότερα. Το πρόγραμμα περιφερειακής ανταπόκρισης, όπως βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια, περιλαμβάνει εννέα εταίρους στις τέσσερις χώρες. Εμείς ζητάμε 810 εκατομμύρια από την διεθνή κοινότητα και ευχαριστούμε τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γενναιότερη βοήθειά τους. Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ ε, λεπτομερό στη διαφάνεια. Ε, ξέρω ότι δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος, αλλά σε γενικές γραμμές αυτές είναι οι βασικές ανάγκες που πρέπει να καλύψουμε. Και θέλω να σας πω ότι το βασικό χαρακτηριστικό των αναγκών μας βλέπουμε είναι ε, τροφή, τρόφιμα, ε, υγεία, διατροφή, εκπαιδεύση και προστασία. Αυτά είναι τα βασικά θέματα. Και βέβαια δεν έχουμε πάρει τους απαραίτητους πόλους ε, που θα θέλαμε. Έχουμε πάρει μόνο ένα ποσοστό του απαιτούμενου ε, ποσού. Αν δεν έχουμε όμως τα απαραίτητα χρήματα, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις υποχρώσεις μας. Και όπως ακούσατε από τη συνάδελφό μου από το Παγκόσμιο ε, Επιστημιστικό Πρόγραμμα, ξέρουμε ότι στην Κένια, στην Ουγκάντα αλλά και στο Νότιο Σουντάν υπάρχουν ε, προγράμματα περικοπής των τροφίμων. Και αυτό λόγω του ότι δεν υπάρχουν χρήματα για κανένα άλλο λόγο. Πάντως υπάρχει ένα πράγμα που αφορά τους πρόσφυγες και είναι το εξής. Μερικές φορές οι πρόσφυγες δεν έχουν ε, αρκετά τρόφιμα και αυτό ε, μπορεί να είναι πηγή συγκρούσεων και τριβών. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Τώρα, εδώ αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσετε η προστασία για μας, για να μπορούμε να απευθυνόμαστε στις κυβερνήσεις, να στηρίζουμε τις τοπικές κυβερνήσεις και βεβαίως να έχουν όλοι κατά νου ότι μιλάμε και για πολλά ασυνόδευτα παιδιά. Περίπου 37.000 ασυνόδευτα παιδιά και σας λέω στις ε, περισσότερες ε, ε, κοινωνίες προσφύγων μιλάμε για γυναίκες και παιδιά. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Τώρα, για το 2015 νομίζω πρέπει να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Αυτές είναι οι μεγάλες προτεραιότητες όσον αφορά τις διάφορες χώρες. Και εδώ υπάρχει κάτι, μια σύμπτωση. Όλοι απαιτούν και θέλουν πρόσβαση σε τρόφιμα, σε νερό, σε παιδεία, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη παιδείας. Στην παιδεία ε, υπάρχει και έλλειψη υποδομής. Θέλουμε να τη βελτιώσουμε την υποδομή, γιατί όπως είπαν και οι συνάδελφοι, η ένοπλη σύγκρουση δεν θα επιληθεί σύντομα και έτσι αυτό που είναι απαραίτητο είναι η εκπαίδευση των παιδιών έτσι ώστε όταν θα επιστρέψουν να είναι χρήσιμοι πολίτες για να βοηθήσουν την κοινωνία. Και αυτό που βλέπουμε από τους πρόσφυγες που έφυγαν πριν από 10 χρόνια, γιατί μερικοί έχουν εκτοπιστεί τρεις φορές. Ένα πράγμα που βλέπουμε είναι ότι μερικοί από αυτούς συνεργάζονται μαζί μας για να βοηθήσουν τους άλλους γιατί εκπαιδεύτηκαν στην Ουγγάντα, στην Κένια, στην Αιθιοπία. Έτσι λοιπόν για μας ε, η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική και έχουμε επενδύσει πάρα πολύ ε, σε αυτούς τους ε, τομείς. Τώρα, επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. πολύ γρήγορα θα αναφερθώ σε συγκεκριμένες χώρες για να αποκτήσετε μία γεύση. Στην Αιτιοπία αυτή τη στιγμή έχουμε 276.000 πρόσφυγες. Περίπου 200.011 από αυτούς εισήλθαν παράνομα στη χώρα. Πάμε τώρα στην Κένια. 46.000 εδώ πρέπει να βελτιωθεί η υποδομή Νότιο Σουδάν το αναφέρω το Νότιο Σουδάν λόγω της κατάστασης των προσφύγων στη χώρα αυτή Σουδάν εδώ είναι η περιοχή που εφέτος ε, δεχτήκαμε πάνω από 80.000 πρόσφυγες στην Ουγκάντα η ροή προσφύγων ήταν λίγο πολύ προβλέψιμη, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι με την κυβέρνηση της Ουγκάντα που εγκατέστησε τους πρόσφυγες όχι σε καταβλισμούς αλλά σε χωριά. Και όσον αφορά την περιφερειακή ανταπόκριση, βλέπετε τι χρειάζεται σε κάθε χώρα. Τα βλέπετε, δεν χρειάζεται να τα διαβάσω, και παρακαλώ στην επόμενη διαφάνεια. Αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΕΚΟ, για την υποστήριξη που μας προσφέρει και να πω ότι κατά την άποψή μας αυτή η κρίση του Νότιου Σουδάν θα διαρκέσει περισσότερο. Γιατί ακόμα και αν αύριο υπήρχε ε, πολιτική λύση, είναι μάλλον απίθανο να αρχίσουν οι πρόσφυγες να διασχίζουν τα σύνορα, κυρίως γιατί όπως σας είπα οι περισσότεροι από αυτούς είναι εκτοπισμένοι ε, δύο και τρεις φορές και οι περιοχές από τις οποίες προέρχονται έχουν καταστραφεί πλήρως. Δεν υπάρχει τίποτα για να επιστρέψουν. Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ πάρα πολύ ενδιαφέροντα τόσα μας είπατε. Βέβαια ήταν και μακροσκελής παρουσίαση και δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ε, πριν αρχίσουμε τη συζήτηση, να δούμε ένα σύντομο βίντεο με τίτλο «Νιάια Story», ιστορία της Νιάια. Από από την αποστολή των Μένων Εθνών στο Νότιο Σουδάν. Υπότιτλοι AUTHORWAVE sen yenge ya ta kan sel gwa mun yur na sun kana na na bel sel gwa mun te na sun dan na yi wa kuma me na kan ba ku dun

άμα το θέλω πως. Σε αμάν δεν νομίζω και εγώ πολύ. Εγώ ζω να μου λέω κάτι. Εγώ δεν λέω να λέω το Uh, Έχουμε τον κύριο Γκερέρο στον ε, κατάλογο των τον πρώτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την παρουσίαση αυτή και όλος ιδιαίτερος θέλω να ευχαριστήσω τις κυρίες Λούμα και Πίτερς και όποιον άλλο προσωπεί οργανώσεις ε, που έχουν επιτόπου ανθρωπιστικά συνεργεία αλλά και όλους όσους εργάζονται βέβαια υποστηριζόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να αναγνωρίσω την προσπάθεια που καταβάλλετε σε τόσο δύσκολες ε, δραματικές συνθήκες, αφόρητες συνθήκες με ψηλό κόστος και μάλιστα και απώλεια ζωής έχουμε, απώλεια ζώων. Μετά από αυτά τα λόγια αναγνώρισης, πρέπει να σας πω ότι τα στοιχεία που μας δώσατε για τα άτομα που είναι υποσυτισμένα, που είναι εκτοπισμένα, μακριά από, την, από τα σπίτια τους, μέσα σε πόλεμο και καθεστώς βίας, αφού είδαμε όλα αυτά τα στοιχεία και είδαμε και αυτό το βίντεο, το εντυπωσιακό αυτό βίντεο, που έχει να κάνει με τη βία κατά των γυναικών συγκεκριμένα και κατά των παιδιών πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα συντομία να σας μεταφερω τεσσερις τέσσερις-πέντε σκέψεις μου. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό το οποίο είπατε κι εσείς, ότι πρόκειται για μια βαθιά ανθρωπιστική κρίση, η οποία προέρχεται από μια ένοπλη σύγκρουση και επομένως ε, έχει ρίζες. Και η λύση μπορεί να βρεθεί μόνο στο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή με την αποκατάσταση της ειρήνης μπορεί να δοθεί λύση. Γιατί μια χώρα ε, που ουσιαστικά μόλις ανεξαρτητοποιήθηκε χωρίς ε, με τρόπο να βλέπουμε πώς αυτό θα μπορούσε να λυθεί γρήγορα ξεκίνησε μια διένεξη, μια αντιπαράθεση που βλέπουμε που καταλήγει. Επίσης πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες για την ε, ειρήνευση στην περιοχή. Και αν ε, έχω σωστές πληροφορίες, την τελευταία φορά που συζητήθηκε το Σουδάν σε Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ήταν το Δεκέμβριο του 2014. Από τότε έχει πέρασει μισός χρόνος. Η κατάσταση επιδεινώθηκε, ο πόλεμος ε, εντείνεται. Μήπως είναι κατάλληλη στιγμή να το ξανασυζητήσουμε σε υψηλό επίπεδο εντός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να λάβουμε μια αποφασιστική δράση σε συνεργασία και με την Αφρικανική Ένωση. Ο κ. Μουντία πάρα πολύ ξεκάθαρα μας ε, απέδειξε ότι έχουμε περιφερειακού χαρακτήρα ε, διένεξη ε, αντιπαράθεση. Δεν περιορίζεται μόνο στο Νότιο Σουδάν και το Σουδάν. Άρα νομίζω ότι η πολιτική εμπλοκή της Αφρικανικής Ένωσης είναι σημαντική, είναι αναγκαία και αποφασιστική. Άρα πρέπει από πολιτικής πλευράς να απευθύνει η έκκληση ίσως και μέσω της ΥΠΑ της εκπροσώπου η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σχέση όπως είπα και με την Αφρικανική Ενότητα και να εργαστούν πάνω στο Δεύτερον, πόροι μας είπατε και μίλησα λίγο πριν κατηδίαν με την ε, κυρία Λούμα, την εκπρόσωπο του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών ε, για το πιστικό πρόγραμμα. Μα είπε ότι τον πρώτο χρόνο κάπω καλύφθηκαν οι ανάγκε σύντηση, αλλά όταν εντάχθηκε ο πόλεμο και όταν είχαμε από το προηγούμενο έτος το δεύτερο τώρα χρόνο είναι αδύνατο να καλυφθούν οι ανάγκες σε τρόφιμα. Για τον επιπλέον λόγο ότι ούτε και η χώρα πλέον δεν είναι σε θέση να παράγει από μόνη της, γιατί οι παραγωγικές ζώνες βρίσκονται μέσα στο μέτωπο, το πολεμικό. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγική διαδικασία. Άλλωστε επιδεινώνεται και το θέμα λόγω των τεχνολογικών εξέλιξεων. Μπορεί δηλαδή να υπήρχε κατάπαυση του πυρός, αλλά επειδή έρχονται οι βροχές πάλι δεν ε, μπορεί να γίνει αυτό και άρα συνεχίζονται και οι μάχες. Τώρα, τρίτον, εκπαίδευση και UNICEF. Όπως ξέρουν όλα τα μέλη της Επιτροπής μας, αυτή η Επιτροπή εδώ έχει ε, δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην πρόθεση της εκπαίδευσης των παιδιών σε χώρες που βιώνουν ανθρωπιστική κρίση και βρίσκονται και σε εμπόλεμη κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν και θα αναλάβουμε διάφορες πρωτοβουλίες για να διατεθούν περισσότεροι πόροι στην εκπαίδευση των παιδιών σε αυτό το περιβάλλον κρίσης. Και υπογραμμίζω και εγώ αυτό που επισήμανε η πρόσωπος ε, της UNICEF, η Πίτερς. Δηλαδή ότι συσσωρεύονται οι ανάγκες για τον τομέα αυτό, στον τομέα της παιδείας. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω κάτι το οποίο, για το οποίο ενημερώθηκα από μια οργάνωση η οποία εργάζεται επί τόπου, ότι δηλαδή πρέπει να διευρεθεί η έννοια περί περιοχών προτεραιότητας. Όταν έχουμε σπάνιδα πόρων, σίγουρα είναι λογικό ότι εστιάζουμε εκεί όπου θεωρούμε ότι θα χρειαστεί περισσότερο από τις άλλες να εστιάσουμε. Μέχρι τώρα οι χρηματοδότες εστίασαν στο Unity, Απερνάλ και Τζογκλέι, σε αυτές τις πολιτείες. Αν όμως είναι οι πληροφορίες που έχω σωστές, υπάρχει επέκταση της σύραξης και καλό είναι να επεκταθεί βοήθεια και να μην περιοριστεί μόνο σε αυτές τις περιοχές. και επειδή πάντα είμαστε υπέρ της ε, συσχέτισης ανθρωπιστικής βοήθειας με την αναπτυξιακή, θα ήθελα να ζητήσω τον κύριο Ντεμπρόι αν και σε ποιο βαθμό ΕΚΟ και ΝΤΕΦΚΟ συνεργάζονται για να δώσουν απάντηση στην κρίση. Thank you. Mr. Ευχαριστούμε. Τσέλερ πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τον Νότιο Σουδάν. Και δυστυχώς δεν μας φέρατε καλύτερα νέα, πιο χαρμόσυνα νέα από αυτά που είχαμε ακούσει στο παρελθόν. Από ό,τι φαίνεται επιδεινώνεται η κατάσταση στο Νότιο Σουδάν. Οξύνεται θα έλεγα η βία. Εγώ τον Ιανουάριο είχα πάει στη χώρα στα πλαίσια μιας αποστολής επιτήρησης εκλογών και είδα πραγματικά εκεί ποιε ήταν οι προσδοκίες του τοπικού πληθυσμού. Οι άνθρωποι προφανώ ήταν υπέρ της ανεξαρτησία της χώρας τους αλλά συνειδητοποίησαν ότι έρχονταν δύσκολοι καιροί. Συντοπίσαν ότι η σύγκρουση δεν θα ήταν μεταξύ του Βορρά και του Νότου, αλλά θα υπήρχε τελικά ένα εμφύλιος φόλεμο ο οποίο θα ξεσπούσε στη χώρα αυτή και ο οποίο τελικά θα έπλητε σχεδόν το σύνολο της χώρας. Και βλέπουμε ότι τελικά αυτό επιβεβαιώνεται. Και συνειδητοποιούμε τώρα ότι η μόνη πόρη της χώρας είναι κάποια αποθέματα πετρελαίου στο βόρειο τμήμα της χώρας. Αλλά ακόμα και η παραγωγή αυτή έχει σταματήσει. Οι εταιρείε που είχαμε εκεί πέρα στο παρελθόν τελικά αποχωρούν όλο και περισσότερο επειδή δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια του προσωπικού του Και αν λάβουμε υπόψη μα και όλα αυτά τα οποία μας είπατε για τι ροέ προσφύγων, όχι μόνο στο εσωτερικό τη χώρα, αλλά και στι όμορε χώρε, τότε συνειδητοποιούμε ότι η κατάσταση όλο και θα επιδεινώνεται, η βία και οι συγκρούσει θα απλώνονται όλο και περισσότερο. Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή στο άμεσο μέλλον μια κάποια κεχηρία και οπότε είχαμε απόπειρα και στο παρελθόν, αυτή δεν κράτησε ούτε καν 24 ώρες. Δεδομένης λοιπόν της κατάστασης, θα πρέπει να προσεγγίσουμε την κρίση αυτή με τρόπο εντελώ διαφορετικό. Πρέπει να κάνουμε μία έκκληση προς όλους όσοι δραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή την περιοχή και αν δεν κάνω λάθος τον ε, Ιούνιο απεστάλει ένα συντονιστή των Εθνών στην περιοχή προκειμένου να βοηθήσει τους εμπλεκόμενους στην διένεξη αυτή να καταλήξουν σε μια κεχηρία και από ό,τι φαίνεται εκδιώχθηκε από τη χώρα ο άνθρωπος αυτός. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την κατάσταση. Δεν μπορούμε να έχουμε καμία εμπιστοσύνη ότι επί τόπου υπάρχει μια κάποια πολιτική βούληση προκειμένου να επικρατήσει τελικά ειρήνη. Θεωρώ λοιπόν ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να συντοπίσει ότι δεν μιλάμε πλέον για μια διένεξη που πλήττει τον Νότιο Σουδάν, αλλά και τις όμορες χώρες, όλη την γύρω περιοχή. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να δράσουμε ακριβώς όπως το κάναμε και στην περίπτωση της σύγκρουσης της Ουκρανίας. Δηλαδή εκεί παγώσαμε τους λογαριασμούς, απαγορεύσαμε την είσοδο Αυτά είναι κάποια μέτρα. Διάβασα ότι υπάρχουν περίπου 14.000 κιανόκρανοι των Ηνωμένων Εθνών στο Νότιο Σουδάν. Ε, άρα δηλαδή και αυτοί θα πρέπει κάτι να κάνουν για να αποτρέψουν ε, το χειρότερο. Μπας περιπτώσει, όπως ήδη σας είπα, με λόγια και μόνο δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στο Νότιο Σουντάν. Χρειαζόμαστε πιο ριζικά μέτρα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ύπατη εκπρόσωπος και τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να δραστηριοποιηθούν, να λάβουν πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, συνεχίζω σε αυτά που μόλις τώρα είπε ο συνάδελφος και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι το θέμα των κυρώσεων. Ε, δεν είναι δυνατόν ε, να επιτρέπουμε σε κάποιους αξιωματικούς να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς τους. Αυτή εντάξει μπορούμε να τους συμμορήσουμε αλλά να είναι πιο ε, αυστηρές οι κυρώσεις. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να τιμωρηθούν, αλλά οι κυρώσεις πρέπει να αφορούν το κράτος. Βλέπουμε ότι τα χωριά συστηματικά καίγονται, έχουμε μπρισμούς, εξαντραποδισμούς, άρα δηλαδή πρέπει να δούμε λιγάκι πού ακριβώς ξεκινάει αυτή η αλυσίδα. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δούμε το κράτος. Αυτή είναι η ε, κορυφή, η αιχμή του προβλήματος. Και εφόσον μιλάμε για κυρώσεις, ε, πρέπει να προσέξουμε να επιβάλλουμε τις σωστές κυρώσεις. Και θέλω να σας πω, είμαι πεπισμένη ότι πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο από ό,τι το είχαμε συνηθίσει. Αν πραγματικά θέλουμε να σταματήσουμε αυτή την εξατλίωση. Βεβαίως και η ανθρωπιστική βοήθεια είναι σημαντική, είναι σημαντική αλλά και εσείς οι ίδιοι το είπατε πόσο δύσκολο είναι να γίνει κάτι, όχι μόνο γιατί λείπουν τα χρήματα και αυτό είναι ντροπή, αλλά και να υπάρχουν πολλά δεν μπορούν να γίνουν. Και έχω ερωτήσεις. Φτάνει ε, να στείλουμε και ανόκρανους ε, παραδείγματος χάρη για να ε, διασφαλίσουμε τις οδούς διαφυγής ή τι πρέπει να γίνει για να προσφέρουμε προστασία. Δεν λέω στρατιωτική επέμβαση, αυτό είναι το τελευταίο που μπορεί να γίνει. Αλλά για να δρομολογηθεί διαδικασία ειρήνης νομίζω ότι και πέρα από τις ειρηνευτικές ε, διαπραγματεύσεις πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις ε, ε, επιτόπου στους Σουδανούς και ίσως και εμπαργό όπλων και αυτό πρέπει να το τηρούν όλοι να μην το παραβιάζει κανείς ούτε και η Ρωσία να ισχύει για όλους γιατί αλλιώς πώς να ε, μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση αν από παντού ε, έρχονται όπλα ή αν όχι όπλα πυρομαχικά. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε και όχι να περιστούμε στις συζητήσεις αλλά να περάσουμε και στην πράξη. Και σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για τη βοήθεια που παρέχετε επί τόπου. Πριν δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες, θα ήθελα να ρωτήσω αν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράσης εκπροσωπείται και θέλει το λόγο. Κυρία Νίπολ, κάπω έτσι. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτά τα οποία ακούω εδώ ευθυγραμμίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις δραστηριότητες ε, τη ΥΠΑ εκπροσώπου, που συνεργάζεται πολύ στενά με τους ε, δύο επιτρόπους, Τηλιανίδη και Μίμητσα. Και μάλιστα εγώ προσωπικά συνόδευσα τον Επίτροπο στην επισκέψή του στο Νότιο Σουδάν, διότι θεωρούμε ότι είναι μια καταστροφή που μας αφορά όλους από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Και όπως πολύ σωστά λέτε, Πραγματικά βλέπουμε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει καθόλου ισχυρή βούληση από καμία από τις πλευρές για εξέβρεση πολιτικής λύσης και αυτό το συμπεριλάβαμε στην δήλωσή μας, η οποία δημοσιοποιήθηκε επευκαιρία της επαιτίου της ανεξαρτησίας νωρίτερα αυτό το μήνα. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση, διότι και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να, να κερδίσουν με τη στρατιωτική δράση. Πάνω από ένα χρόνο έχουμε διαμεσολάβηση, την οποία υποστηρίξαμε επειδή θεωρούσαμε ότι στην περιοχή ε, πρέπει, από την περιοχή πρέπει να ξεκινήσει αυτή η διαμεσολάβηση και κυρίως από την Ουγκάντα και από το Σουδάν που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο γιατί έχουν ε, και ζωτικά συμφέροντα στη χώρα, στο Νότιο Σουδάν δηλαδή. Έχουμε και τον ειδικό εκπρόσωπο για το κέρας Αφρικής, ε, τον Αλέξανδρο Ρόντο, ο οποίος τους τελευταίους μήνες πολύ μεγάλο μέρος που έχει περάσει στο Νότιο Σουδάν και συνεργάζεται και αυτός με τους επεσταλμένους ε, της Νορβηγίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και τον ΙΠΑ, παρακολουθώντας ε, και με την ΙΓΑΝΤ αυτή την ε, κατάσταση. Να πω ότι και άλλες χώρες πρέπει να στηρίξουν την ΙΓΑΝΤ. Έχουμε τη μεσολάβηση της ΙΓΑΤ που ούτε όμως και αυτή απέφερε καρπούς όπως γνωρίζουμε. Μόλις ο ΙΕ ενέκρινε κυρώσεις, όπως είπατε και εσείς, για έξι στρατιωτικούς ηγέτες, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε επιβάλει ήδη νωρίτερα κυρώσεις. Η συζήτηση για την επέκταση αυτών των κυρώσεων συνεχίζεται στο Συμβούλιο και στην Τζούμπα και εδώ στις Βρυξέλλες έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό και τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Υπάρχει βέβαια και απόψη ότι θα πρέπει τις κυρώσεις να τις υποστηρίξει και η περιοχή γιατί οι λογαριασμοί ε, των ηγετών είναι πιο πολύ στην περιοχή παρά εδώ. Δύσκολα μπορεί κανείς να στοχεύσει στους ηγέτες, ε, τους προτεργάτες όλης αυτής της σύγκρουσης, αν δεν έχει τη στήριξη της σύγκαντα. Αλλά είναι μια δύσκολη συζήτηση, είναι σε εξέλιξη. Είπατε εκπρόσωπος παρακολουθεί εκ του σύνεγγης ε, το θέμα. Διότι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ασκηθούν περισσότερες πιέσεις. Η λύση πρέπει να είναι πολιτική. Μόνο έτσι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια βιώσιμη λύση. Συνεργαζόμαστε στενά με την Ίγκα, την Αφρικανική Ένωση και βέβαια και με τα Ηνωμένα Έθνη. Υπάρχει ε, όπλων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, εφαρμοζόταν στο Σουδάν όταν ήταν ένα κράτος. Αυτό το εμπάργκο μεταφέρθηκε αυτόματα και στο Νότιο Σουδάν. Υπάρχει, μάλλον είναι εμπάργκο της Ένωσης και του Ηνωμένων Εθνών. Okay, uh, Τρία λεπτά ο καθένα σας αρκούν για να απαντήσετε. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Ντεμπράουερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολλά από τα ερωτήματα αφορούσαν την ΕΕΔ και δεν, να μπορώ παρά να συμφωνήσω πλήρω με την Κλόντια. Ο κύριο Τηλιανίδη πράγματι ε, γύρισε από την περιοχή πεπισμένος ότι θα πρέπει να ε, κάνουμε κάτι με τις κυρώσεις. Ε, το Συμβουλίο Ασφαλείας έκανε πρώτο κυρώσεις, θεωρήθηκε από τον πρόεδρο και ως άστοχο, άστοχη κίνηση και θεωρώ ότι είναι σωστή αυτή, αυτός ο χαρακτηρισμός ε, δεν ήταν ε, σωστά στοχευμένες οι Επίσης υπήρχε και το δεχόμενο ενός εμπάργκο όπλων. Ε, τίθεται και θέμα τέτοιο στη, ε, στους, στα Έθνη και ίσως υπάρχει λύση και σε αυτό. Τώρα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μας με, το γάμα δέλτα, με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ανάπτυξη, εξαιρετική είναι η συνεργασία μας, εκπροσωπείται στην αίθουσα η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ αυτή. Βέβαια Πρέπει να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Νότιο Σουδά που δεν έχουμε καταφέρει βέβαια να έχουμε το LRD, την All Residents Approach, να την υιοθετήσουμε εντελώ δεν έχουμε καταφέρει. Είπε και η κυρία Λούμα πράγματα ε, αποτροπιαστικά. Πρέπει να δείτε τι κάνουν ε, τα συνεργεία εκεί των ανθρωπιστικών οργανώσεων, ε, γιατί χάρη σε αυτά γίνεται κάτι. Αλλά πρέπει να δούμε τα κατεπήγοντα ζητήματα πρώτα και μετά θα έχουμε επαφές και συνεργασία και με τους άλλους φορείς. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε πρώτα τα κατεπήγοντα, τις κατεπήγουσες ανάγκες και έπειτα να δημιουργήσουμε ένα είδος αντοχής, αντίσταση και να δημιουργήσουμε και ένα κλίμα συμφιλιωτικό. Αν ποτέ δηλαδή υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για να συμφιλειωθούν πλευρές κάτι που δεν το ανέφερα διεξοδικά. Συνεπία της σύγκρουσης αυτής είναι και η οικονομική ύφεση. Καταραίει στη γεωλεξία το Νότιο Σουδάν. Μεγάλη πτώση, ε, βουτιά κάνει το εθνικό νόμισμα, όπως να τα πει καλύτερα κάποιος από τους άλλους εδώ στο πάνελ. Οι τιμές των τροφίμων ή των αγαθών είναι ε, πάρα πολύ υψηλές. Ε, μέχρι και το νερό, ένα μπουκάλι νερό, τα καύσιμα ε, είναι απλησίαστα για τους πολίτες λόγω των τιμών πράγματι ήταν πρόβλημα για κάποιες πολιτείες, αναφέρατε κάποιες, αλλά τώρα διευρύνει την κρίση και για την ίδια την Τζούμα γίνεται πλέον ε, πρόβλημα. Έχουμε ε, επιδίνωση και ίσως έχει ως αποτέλεσμα την επιδίνωση της πολιτικής κρίσης αλλά και την ε, όξυνση της οικονομικής κρίσης ε, λόγω αυτών των ε, επεισοδίων και της βίας. Εμείς είμαστε παρόντες σε όσο να το περιοχές της χώρας μπορούμε. Τα κριτήρια παρέμβαση χορηγία για μα είναι ε, η ευαλωτότητα, όπως γνωρίζετε, και τα παιδιά. Ο Επίτροπο Τηλιανίδη ε, προσωπικά προσδίδει στην προστασία και την εκπαίδευση των παιδιών την ύψιστη δυνατή προτεραιότητα. Και το Νότιο Σουδάν είναι το καλύτερο δυνατό, όχι βέβαια, πώς να το πω, ε, ήθελα να πω τέλος ότι είναι ακριβώς ο τόπος στον οποίο μπορούμε να δράσουμε πάνω σε αυτό το, ε, σε αυτό το μέτωπο. Εμείς πάντως σας ευχαριστούμε πολύ για τη δική σας υποστήριξη και σταματώ εδώ. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. κυρία Λούμε, έχει τώρα το λόγο. Συμφωνώ. Συμφωνώ ότι η ε, λύση στην κρίση που αντιμετωπίζουμε στο Νότιο Σουδάν μπορεί να είναι μόνο πολιτική. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμο. Μία παρατήρηση όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα. Και εκεί έχουμε πολύ σημαντική κρίση και εκεί πρέπει να κάνουμε κάθε το δυνατό προκειμένου να επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε δεν υπάρχει πραγματικά καμία απόλυτο ελπίδα. Τα παιδιά αυτά θα καταλήξουν σε παραστροτικέ οργανώσει και ήδη είναι πολλές οι οργανώσεις αυτές οι οποίες θα συνεχίσουν να στρατολογούν παιδιά και θα συνεχίσουν και θα διονύσουν τον πόλεμο. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα λοιπόν για τη χώρα αν δεν υποστηρίξουμε το εκπαιδευτικό σύστημα. Όσον αφορά τώρα την μακροοικονομική κατάσταση στο Νότιο Σουδάν. Έχουμε μια οικονομία η οποία παράγει ένα και μοναδικό προϊόν, το πετρέλαιο, τίποτα παραπάνω. Ξέρουμε βέβαια ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η παραγωγή εξαιτία του πολέμου αλλά έχουν μειωθεί ούτως ή άλλως παγκοσμίω και οι τιμέ του πετρελαίου. Και κατά συνέπεια ο προπολογισμό της χώρας έχει μειωθεί πάρα πολύ. 300 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό το οποίο χρειάζεται η χώρα για τον προπολογισμό της και προφανώς ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτού του προπολογισμού καταφέρνει αυτή τη στιγμή να παράγει και ήδη ένα εκατομμύριο πηγαίνει σε αμυντικές δαπάνες και καθόλου χρήματα δεν πηγαίνουν στις κοινωνικές υπηρεσίες. Επίσης έχει υποτιμηθεί πάρα πολύ το εθνικό νόμισμα όπως είπατε με αποτέλεσμα να αυξάνονται πάρα πολύ τιμές βασικών προϊόντων, καύσιμα, εφιαλωμένο νερό, ψωμί κτλ. Και πάρα πολλοί απαιτούν αυτή τη στιγμή ότι ακόμα και τα βασικά αυτά προϊόντα θα πρέπει να πληρώνονται σε αμερικανικά δολάρια καταλαβαίνετε ότι κατά αυτόν τον τρόπο ασκείται ιδιαίτερη πίεση στον πληθυσμό και αυξάνεται πάρα πολύ η κλιματική δραστηριότητα στην Νότιο Σουδάν. Πράγμα το οποίο με τη σειρά του δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη ζωή των πολιτών. Ξέρετε ότι ακόμα και οι επιτόπου εργαζόμενοι για τα ανθρωπιστικά προγράμματα φοβούνται πλέον για τη ζωή τους. Δεν μπορούν να κάνουν με ασφάλεια τη δουλειά τους. Ενώ ανησυχούμε για τον πληθυσμό στην Ήπεθρο, όπω είπατε εσεί, αρχίζουμε και ανησυχούμε όλο περισσότερο για τον αστικό πληθυσμό, καθότι και οι πόλεις πλέον πλήττονται από, την, από τον πόλεμο και υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι που πλήττονται από υποσυτισμό ακόμα και στι πόλει πλέον. Η μακροοικονομική λοιπόν εικόνα τη χώρα δεν έχει να κάνει μόνο με την επιστηστική ανασφάλεια, πλήττονται και άλλοι τομεί. Αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου ο υγειονομικό τομέα πλήττεται πάρα πολύ. Πολύ σύντομα δεν θα έχουμε φάρμακα στη χώρα. Αν δεν γίνει κάτι μέχρι τον Νοέμβριο, η χώρα δεν θα έχει τα απαραίτητα βασικά φάρμακα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δίνουμε μία μάχη όχι μόνο κατά της ε, επιστηστικής ανασφάλειας, αλλά κατά μιας ε, ευρείας υγειονομικής κρίσης που πλήττει το σύνολο της χώρας. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πίτερς, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις σας. Συμφωνούμε και εμείς ότι η λύση θα πρέπει να είναι σαφώς πολιτική, ωστόσο θα θέλαμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Προτεραιότητά μας είναι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε οργανισμούς όπως τον δικό μου προκειμένου να επιτηρούμε όλα τα φαινόμενα βίας κατά των παιδιών και των γυναικών. Η χρηματοδότηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάτι τέτοιο. Χρειάζεται όμως και πολιτική υποστήριξη προκειμένου να καταδικάσουμε αυτές τις πρόδειλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παιδιών και γυναικών. Ευχαριστούμε λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και την ύπατη εκπρόσωπο για τη δήλωσή της που έκανε κατά την τέταρτη επέτειο της ανεξαρτησίας του Νοτιού Σουδάν. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες. Είναι πραγματικά παράδεκτο οι φρικαλαιότητες, η βαναυσότα να συνεχίσει στη χώρα αυτή χωρίς να υπάρχει καμία καταγγελία σε πλήρες καθεστώς ατιμορρησίας. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι διεθνείς οργανισμοί να συνεχίσουν να παρακολουθούν τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών, των γυναικών και των κοριτσιών. Όσον αφορά την υποστήριξη για το σύστημα παιδείας, συμφωνούμε και εμείς, με έχει καλύψει η συνάδελφος, δεν θα πρέπει μόνο να υποστηρίξουμε Κάποια παιδιά, ήδη 400.000 παιδιά κατάφεραν να επιστρέψουν στο σχολείο, παρόλα αυτά εκατομμύρια παιδιά παραμένουν εκτός σχολείου. Πολλά από τα παιδιά αυτά είναι νέοι έφηβοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η μοίρα των παιδιών αυτών, όχι μόνο στο Νότιο Σουδάν, αλλά και στις όμερες χώρες. Είναι έρμεο των, α, α, της στρατολόγησης που γίνεται από παραστρατιωτικές οργανώσεις. Οφείλουμε λοιπόν να αρχίσουμε να επενδύουμε προκειμένου να επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο. Συμφωνώ με τον κύριο Ντεπάουερ ότι ε, υπάρχει ήδη ένας πολύ επικοδομητικός διάλογος επιτόπου αλλά και στα θεσμικά όργανα στι Βρυξέλλες με την ΤΕΦΚΟ και την ΕΚΟ, τις δύο δηλαδή γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει όμως να δούμε πώς θα καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε περισσότερο την εκπαίδευση. Χρειάζονται τεράστιε επενδύσει όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα και οι επενδύσεις αυτέ δεν μπορούν να έρθουν μόνο από τα κονδύλια ανθρωπιστική βοήθεια. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα των κυρώσεων να τονίσω ότι κάθε φορά που επιβάλλουμε κυρώσει σε μια χώρα θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι θα πρέπει να υπάρχουν και τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για να προστατευτούν τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού, γιατί πολύ συχνά όταν επιβάλλουμε κυρώσει, οι πρώτοι που πλήττονται είναι οι γυναίκε και τα παιδιά. Και έχουμε πάρα πολλέ αποδείξει για το φαινόμενο αυτό σε πάρα πολλέ χώρε. Σα ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πίτερ. Δεν αναλώσατε όλο το χρόνο που σα αναλογούσε. Ο κύριο Μούντια τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά να τονίσω και εγώ κάποια πράγματα που είπαν οι προλύσαντες. Ας δούμε όμως και την περιφερειακή διάσταση. Στις περισσότερες χώρες που έχουμε τέτοια πολύ, μεγάλα, πολύ μεγάλες ομάδες προσφύγων, αυτό το οποίο βλέπουμε, είτε μιλάμε για την Ουγκάντα, είτε μιλάμε για την Κένια ή για τον Νότιο Σουδάν, σε κάθε περίπτωση έχουν καταβληθεί προσπάθειες από τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να παραχθούν γενομικές να παρασχεθούν με συγχωρείτε γενομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες στα πλαίσια του τομέα της εκπαίδευσης. Το πρόβλημα όμως με τις ε, περιοχές αυτές που φιλοξενούν ε, πολύ μεγάλους αριθμούς προσφύγων είναι ότι τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Στην Κουκούμα για παράδειγμα είχαμε τάξεις που είχαν 40 μαθητές στο παρελθόν Τώρα οι μαθητές αυτοί έχουν γίνει 80 και άνω. Στην Αιθιοπία υπάρχουν πάλι παιδιά τα οποία έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά το σύστημα το ίδιο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, καθότι οι πρόσφυγες είναι πάρα πολλοί. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όχι μόνο να υποστηρίξουμε χώρες και κυβερνήσεις, αλλά τοπικές κοινότητες και περιφέρειες που δέχονται, φιλοξενούν τεράστιο αριθμό προσφύγων. Αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, νομίζω ότι δυσχεραίνουμε την κατάσταση και δεν βοηθούμε το, έργο των τοπικών κυβερνήσεων. Όσον αφορά τώρα τις κυρώσεις, ναι, μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις, αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε και με κάποιες από τις χώρες περιφέρειας αυτής που θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά τον Νότιο Σουδάνα. Ακόμα και αν επιβάλλεται κυρώσεις, όπως είπε και η προαλήσασα, οι κυρώσεις αυτές πολλές φορές δεν έχουν ε, κάποιο άμεσο αντίκτυπο. Αυτό που βλέπουμε πολλές φορές είναι ότι ε, ορισμένοι τελικά παίρνουν τα χρήματά τους, τα κρύβουν κάτω από το στρώμα τους ή πλήττονται τελικά οι πιο ευάλωτοι στις χώρες αυτές. Άλλοι καταφέρνουν να καταφύγουν, οι πιο δυνατοί δηλαδή και οι πιο πλούσιοι μπορούν να πάνε σε άλλες χώρες. Πρέπει λοιπόν να επιβάλλουμε κυρώσεις οι οποίες όμως να είναι πιο ευφυείς και πιο αποτελεσματικές, να μην είναι κλασικές, σύνηθες κυρώσεις. Και έχουμε και ορισμένε χώρες στην όλη αυτή περιοχή που έχουν πολύ σημαντικά συμφέροντα και μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική κατάσταση. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε μία ισότιμη κατανομή της ευθύνης και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Προετοιμαζόμενος για τη συνεδρίαση αυτή, προσπαθούσα να δω πραγματικά ποιες είναι οι περιφέρειες αυτές οι οποίες έχουν εμποδίσει την επίτευξη συμφωνία στο Νότιο Σουδάν. Αν δούμε τις περιφέρειες αυτές θα συνειδητοποιήσουμε ότι ορισμένες έχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα και γι' αυτό το λόγο δεν υπέγραψαν την επιθυμητή αυτή συμφωνία ειρήνευσης. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει προφανώς να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να βοηθήσει τα πράγματα, να επιβάλλει ενδεχομένως κυρώσεις, αλλά θα πρέπει πραγματικά οι υπεύθυνοι αυτοί να βρεθούν περισσότερο στο στόχαστρο των κυρώσεων διότι αν δεν καταφέρουμε να κάνουμε αυτή την εξειδίκευση, αν θέλετε, στις κυρώσεις, πλήττονται και πολλά άλλα τμήματα του πληθυσμού και πολλές άλλες περιοχές εντός και εκτός Νοτιού Σουδάν. Αλλάζει και η ίδια η περιφερειακή διάσταση όμως της ένοπλης αυτής σύγκρουσης στον Νίγηρα, Προτού ξεκινήσει η ένοπλη σύραξη τον Δεκέμβριο, ξέρετε ότι υπήρξε μία αρχή αντιπαράθεση η οποία από περιφερειακή έγινε στη συνέχεια στρατιωτική και πήρε πολύ μεγαλύτερες και διαστάσεις. Βλέπετε ότι και στο Νότιο Σουδάν έχουν αρχίσει να επηρεάζονται και να αποσταθεροποιούνται περιοχές οι οποίες εξ αρχής δεν είχαν εμπλακεί στην ένοπλη σύγκρουση. Και είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι μία ή άλλη περιφέρεια βρίσκεται υπό τον απόλυτο έλεγχο του ενός ή του άλλου στρατιωτικού αρχηγού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η δική μας η δράση, αν δεν στοχεύσει σε συγκεκριμένους στόχους, θα καταλήξει να γίνεται όλο και πιο δαπανηρή, κυρίως όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους, λέει ο Πρόεδρος. Ήταν εξαιρετικές οι παρουσιάσεις σας και ιδιαίτερα χρήσιμη για μας η συζήτηση αυτή που είχαμε. Εξ λοιπόν της Επιτροπής μου σας ευχαριστώ και προφανώς θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το καταπληκτικό σας έργο. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 13, ώρα των ερωτήσεων. Δεν έχουμε λάβει καμία ερώτηση όμως για τη σημερινή μας συνεδρία. Περνάμε στα διάφορα. Θέλετε να θίξετε κάποιο ζήτημα στο σημείο 14, διάφορα. Όχι. Προσεχή συνεδριάσεις. Θα συνεδριάσουμε λοιπόν στις 3 Σεπτεμβρίου και κατά αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνω τη σημερινή μας συνεδρίαση και την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας πριν τις τερινές διακοπές να σε ευχηθώ ένα ηλιόλουστες και ευχάριστες διακοπές. Σας δω το Σεπτέμβριο.